So, Kolleginnen und Kollegen, können wir... Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Τι, τι πάει να πει όχι. Θα ξεκινήσω παρόλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σήμερα το πρωί είχαμε πει γιατί το γράμμα για το, για το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση λοιπόν αναβάλλεται. Αλλά θα περάσουμε στο 9 και πάμε στην ψηφοφορία τώρα. Είστε όλοι έτοιμοι? Α, να και εγώ. έτοιμος. Να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία για την πρώτη παράγραφο. Ψηφίζουμε το συμβαστικό κείμενο με τη συμπλήρωση από το ECR. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται με αυτήν τη συμπλήρωση. Ε, ερώτημα 1. Να ψηφίσουμε το συμβαστικό κείμενο. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Εγκρίνεται. Ερώτημα 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ωραία, να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε για το ερώτημα 2. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, ερώτηση 2α. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ερώτημα 3. Α, συγγνώμη, το δεύτερο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα πρέπει και αυτό να το ψηφίσουμε. Υπέρ κατά. Λοιπόν, να ελέγξουμε. Ψηφίσουμε για το 3, λοιπόν. Το δεύτερο τμήμα. Του 2, λέει τώρα ο πρόεδρος. Ψηφίσατε όλοι. Ναι. Απορρίπτεται. Δεν λειτουργεί κάποιο μηχάνημα. Α, ναι, είσαι κατά, μάλιστα. Απορρίπτεται. Οπότε δεν πειράζει. Ερώτηση 3. Συμβαστικό κείμενο υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές υπέρ. Εγκρίθηκε. Ερώτηση 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 4α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε πράγμα στην τελική ψηφοφορία για την προφορική ερώτηση υπέρ κατά Λοιπόν, εμπάσχευτος, θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ. Παρακαλώ και πάλι η καταληκτική ψηφοφορία για την προφορική αυτή ερώτηση ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ωραία 43 ε, υπέρ, μία κατά, τέσσερις αποχές. Εγκρίνεται η προφορική αυτή ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να κάνουμε μία σύντομη διακοπή για να έρθουν οι εκπρόσωποι των ορισμών και φορέων και να έχουν δυνατότητα να καθίσουν. So, dann ich den Tagesordnungspunkt. Ωραία. Περνάμε στα σημεία 10 έως 13 της ημερήσιας διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων με, τις, με τους τέσσερις οργανισμούς για τους οποίους είμαστε αρμόδιοι εμείς. Προσκαλέσαμε, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, τέσσερις εκπροσώπους των οργανισμών αυτών για να μας πούνε τις δικές τους παρατηρήσεις, τις εμπειρίες που έχουν συλλέξει Καλωσορίζω λοιπόν την Κρίστα Σέντλατσεκ, Διευθύντρια του ΩΣΑ, τον Μάντλεν Σέρμπαν από το Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τον Τζέιμς Καλέχα από το Σεντεφόπ και τον Χουάν Μενέντες Βαλντές, Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ. Δεν θέλω να μακρηγορήσω για να μην φάω το χρόνο σας. Μετά από τις παρουσιάσεις σας θα ξεκινήσουμε συζήτηση με, τους, ε, με τις πολιτικές ομάδες, με τους συντονιστές και νομίζω ότι θα έχουμε αρκετό χρόνο αμέσως μετά για να κάνουμε μια συζήτηση. Πρώτα την κυρία Κρίστα Σέντλατσεκ θα ήθελα να ζητήσω να μας μιλήσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να σας παρουσιάσω τα επιτεύγματα 2015 και ε, στη συνέχεια κάποια ε, σημαντικά θέματα για το 2016. Ξέρετε ότι ο ΩΣΑ ή το σχέδιο εργασιών του οργανισμού βασίζεται ε, στο στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί εκεί έχουμε σημαντικό ρόλο σε πολλούς τομείς αυτού του πλαισίου. Να ξεκινήσω με μία από τις εμβληματικές μας πρωτοβουλίες που είναι η υγεία στον χώρο εργασίας 2014-2015, μια διετής εκστρατεία για, τα, για τις επαγγελματικές ασθένειες και τις ψυχοκοινωνικές ασθένειες στον χώρο εργασίας. Είναι πρόβλημα που αυξάνεται τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργαδότες όλη την Ένωση. Μπορούμε να πούμε ότι περίπου 50% των εργαζομένων αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν στρες στην εργασία τους. Από την άλλη το επαγγελματικό στρες ε, συμβάλλει στην απουσία από την εργασία και την ε, μείωση της ε, παραγωγικότητας και εκατοντάδες μέρες που, χαμένες κάθε χρόνο. Ξέρουμε ότι πολλοί διευθυντές στην Ευρωπαϊκή Ένωση λένε ότι γνωρίζουν το πρόβλημα αλλά μόνο 30% των εταιριών λαμβάνουν μέτρα. Αυτό σημαίνει και αυτή είναι και η δική μας βάση ε, για την διοργάνωση αυτής της διετούς εκστρατείας και στη διάρκεια αυτής της εκστρατείας υποστηρίζουμε όλα τα κράτη-μέλη μέσα από υλικό, μέσα από παρουσιάσεις στα μίντια στις 24 επίσημες γλώσσες της Ένωσης και έχουμε και μια σειρά από δραστηριότητες στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Για πρώτη φορά Συντάξαμε και έναν ηλεκτρονικό οδηγό με στόχο να βοηθηθούν οι μικρές και πολύ μικρές ε, επιχειρήσεις να διαχειριστούν το στρες στον χώρο εργασίας και το βασικό μήνυμα στη διάρκεια αυτών των δύο ετών αλλά και μετά είναι ότι είναι εφικτό να αξιολογηθεί το στρες και η ψυχοκοινωνική πίεση στην δουλειά και υπάρχουν μέτρα που μπορούν να ληφθούν. Γι' αυτό το λόγο παρουσιάζουμε ε, ε, εταιρείε οι οποίες ανέλαβαν θετικά μέτρα για τη διαχείριση του στρες. Στέφτηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η συγκεκριμένη οργάνωση, διοργάνωση στο πλαίσιο της ε, εκστατείας αυτής η οποία ολοκληρώθηκε στις 30 Νοεμβρίου στο Μπιλμπάου. Ένα άλλο πρόγραμμα, κάτι που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερος εσάς, το Κοινοβούλιο, γιατί εσείς αναθέσατε το έργο αυτό στην, στον οργανισμό μας, είναι ε, η πρωτοβουλία για την ε, ε, γύρανση του πληθυσμού και την ασφάλεια και υγεία στον χώρο εργασίας. Εμείς βασιζόμαστε στο έργο που έχει γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο συνολικός στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι να βοηθήσουμε να ενημερωθούν οι φορείς χάραξης πολιτικής, να υποστηρίξουμε την υγεία και ασφάλεια για όλους τους εργαζομένους, να αντλήσουμε διδάγματα για το τι είναι καλή στρατηγική και ποιες είναι οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται επί του παρόντος και να προσφέρουμε και να εντοπίσουμε βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες στρατηγικές. Όλες οι δημοσιεύσεις αυτές θα δημοσιευθούν ε, και θα κοινοποιηθούν το 2016. Πολύ σύντομα λοιπόν θα λάβετε όλες τις πληροφορίες για το γυράσκον εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέμα το οποίο ερευνήσαμε σε 31 χώρες Γι' αυτό και θα αποτελείται η παρουσίασή μας αυτή από 31 εκθέσεις και αυτή η δραστηριότητα νομίζω ότι θα αποτελέσει σημαντικό τμήμα των πληροφοριών για την επόμενη εκστρατεία για την υγεία στον, ε, στο χώρο εργασίας 2016-2017. Μια άλλη δραστηριότητά μας είναι ε, το επιγραμμικό εργαλείο ε, ανάλυσης κινδύνου που έχουμε αναπτύξει, το ΟΕΡΑ που βοηθά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για να μπορούν να συμμορφώνονται με τους κανόνες ε, υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας και αυτοί οι κανόνες ε, αναφέρονται ρητός στο στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εργαλείο αυτό έχει αναγνωριστεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όσον αφορά τη διευκόλυνση της αξιολόγησης κινδύνου και της προώθησης μιας κουλτούρας πρόληψης, ιδίως για τις μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 2015 ήταν πολύ επιτυχημένη χρονιά, γιατί επιτύχαμε πολλούς από τους στόχους που είχαμε θέσει. Για παράδειγμα, έχουμε πλέον 86 ε, νέα εργαλεία όηρα και τουλάχιστον 30 βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης και επίσης διοργανώσαμε σεμινάρια σε εθνικό επίπεδο για να προωθήσουμε το ΩΕΡΑ. Άλλο ένα εργαλείο δημοσιεύτηκε από τον κλαδικό ε, εταίρο από τον τομέα του αθλητισμού. Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε για το ΟΕΡΑ που διεξήχθη το 2015, η πλειοψηφία των εργαλείων ΟΕΡΑ είχαν κάποια κάποιον ή πολύ σημαντικό αντίκτυπο. Και τα ίδια σχόλια έκανε και το ελεγκτικό συνέδριο που είπε ότι σε μεγάλο βαθμό το όιρα είναι ένα πολύ επιτυχημένο εργαλείο και ε, συνεχάρισαν ε, τον οργανισμό του για την ενεργή του δράση. Επίσης έγινε μια έρευνα για νέους και ανερχόμενους κινδύνους στον χώρο εργασία που διεξήχθη το 2016 σε 36 χώρε, 50.000 επιχειρήσεις ε, αξιολογήθηκαν, τα πορίσματα ε, παρουσιάστηκαν τον Φεβρουάριο του 2015 ε, επί Λετωνικής Προεδρίας και τα πορίσματα αυτά παρουσιάστηκαν στο Κοινοβούλιο τον Ιούνιο. Μπορείτε να βρείτε όλα τα πορίσματα αυτά στο, στο σελίδι μας. Είχαμε και ένα ε, σεμινάρια, είχαμε και σεμινάρια προώθηση σε μια σειρά από χώρε, Εστονία, Δανία, Ολλανδία, Νορβηγία και το 2016 θα γίνουν αντίστοιχα ε, αντίστοιχες παρουσιάσεις ε, σε άλλες χώρες, Γερμανία, Γαλλία και το 2016 επίσης θα συνεργαστούμε με την Eurofound και με την Eurostat. Επομένως, η δεύτερη δευτερογενής ανάλυση που θα γίνει το 2016 και 2017 θα επικεντρωθεί στην διαχείριση όσα και την διαχείριση των ψυχοκοινωνικών ε, προβλημάτων. Αυτά ως προς το 2015. Για το 2016 θα ήθελα να επισημάνω τρία βασικά θέματα. Πρώτον, ε, έναρξη της ε, εκστρατείας για την υγεία στο χώρο εργασίας 2016-2017, υγεία για όλους στον χώρο εργασίας και θα επωφεληθούμε από τα προγράμματα και τις δραστηριότητες που ανέφερα νωρίτερα, από αυτό που μας ε, αναθέσατε εσείς και η Κομισιόν, και στόχος μας είναι να προωθήσουμε την βιώσιμη εργασία με εστίαση σε ζητήματα υγείας και ασφάλεια και σκοπός είναι να ενισχυθεί η ασφάλεια και η υγεία στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συμβολή στην βιώσιμη ανάπτυξη και η προώθηση της υγιούς γύρανσης και θα επισημάνει την, τον σημαντικότατο ρόλο της πρόληψης στη διάρκεια της εργάσιμης ζωής μας. Ε, ζωής μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινάει η πρόληψη όταν κανείς ξεκινά την εργασία του. Και σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε υλικό σε όλες τις γλώσσες, θα συνεργαστούμε με όλα τα κράτη-μέλη και για άλλη μια φορά θα ε, αναπτύξουμε ηλεκτρονικά εργαλεία, διαδικτυακά εργαλεία ε, για να μπορεί κανείς να πλοηγείται και στις πληροφορίες ώστε να μπορεί κανείς να σχηματίζει εικόνα, για το πού βρισκόμαστε ως Ευρώπη και πού θα πάμε τα επόμενα χρόνια. Η έναρξη της εκστρατείας θα γίνει 14 Απριλίου ε, με την Ολλανδική Προεδρία και τον Επίτροπο Τίσεν. Άλλα έργα και προγράμματα ε, αφορούν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπου εργαζόμαστε σε διάφορους τομείς και σε διάφορα επίπεδα. Θα ε, συντάξουμε μια επισκόπηση, μια σύνοψη της κατάστασης των μικρών επιχειρήσεων, τι χρειάζεται για να υπάρχει συμμόρφωση με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας. Το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί το 2018, αλλά θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στους φορείς χάραξης πολιτικής, αλλά και για τους εργοδότες. Και τέλος, ένα άλλο πρόγραμμα, μια δραστηριότητα που ξεκίνησε το 2015 στα τέλη της ε, χρονιάς, σχετίζεται με τις επαγγελματικές ασθένειες. Πληροφορίες για την, ε, για την έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες ε, στην Ευρώπη είναι γενικά παροχημένες και είναι απαραίτητες για να αξιολογεί κανείς τον κίνδυνο. Θα εντοπίσουμε ομάδες εργαζομένων υψηλού κινδύνου και θα ε, ορίσουμε και εδώ προτεραιότητες πρόληψης και μέσω αυτής της δραστηριότητας ο οργανισμός σκοπεύει να βοηθήσει τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους φορείς ε, στην, ε, στον εντοπισμό και τη διάγνωση επαγγελματικών ασθενειών στον χώρο εργασίας να θεσπίσουν μέτρα και να θέσουν προτεραιότητες για την έρευνα. Αυτές, αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το 2018 Αυτά για το 2015 και το 2016 και φέτος παρά το γεγονός ότι έχουμε περικοπή προσωπικού που σημαίνει για τον όσα ένα άτομο λιγότερο το 16 και ένα άτομο λιγότερο το 17 θα προσπαθήσουμε παρόλα αυτά να αναδιοργανώσουμε τις δομές μας προκειμένου να ανταποκριθούμε και να επιτύχουμε τους ε, στόχους που σας παρουσίασα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη παρουσίαση. Τώρα πρέπει να αναγνωρίσω ότι έκανα λάθος και δεν χαιρέτησα 25 εκπροσώπους από την, από την Ένωση Χαλιβουργίας του Λογάν Σοτιέ και μια ομάδα 15 μαθητευομένων μεταφραστών από την DG Trend, τη Γενική Διεύθυνση ε, Μετάφρασης και Εκδόσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήρθαν εδώ για να δούμε πώς ακριβώς χειριζόμεθα την ε, πολυγλωσία. Και τώρα να δώσω το λόγο στον James Κάλεχα για τη δική του παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί σας ε, το έργο που έχουμε επιτελέσει το 2015 και τι προβλέπουμε ε, για το 2016. Εμεί ασχολούμαστε με την επαγγελματική κατάρταση και την αγορά εργασία ε, και εστιαζόμαστε στι δεξιότητε και τα προσόντα. Συνεπώ, εστιαζόμαστε σε όλε τι πτυχέ τη μάθηση για εργασιακού σκοπού. Μέσα στο επόμενο δεκάλεπτο θα σας παρουσιάσω θα σας παρουσιάσω τις απαντήσεις που δίνουμε εμείς τις τέσσερις ερωτήσεις που συχνά θέτουμε στους εαυτούς μας. Το πρώτο είναι σε τι πλαίσιο καλείται κανείς να εργαστεί σήμερα και φυσικά αν κοιτάξει κανείς ε, γύρω του σήμερα βλέπει ότι η αγορά εργασίας ε, βρίσκεται σε διαρκή μεταβολή. Και έτσι η εκπαίδευση πρέπει να ανταποκρίνεται στις αλλαγές της αγοράς εργασίας. Επίσης ε, ε, το εργατικό δυναμικό γυράστηκε όλο και περισσότερο και μέχρι το 2025 ε, οι εργαζόμενοι άνω των 55 ετών ε, θα έχουν αυξηθεί σημαντικά. Έτσι λοιπόν εμείς σκοπό έχουμε να εργαστούμε για μια αγορά εργασίας η οποία επίσης θα είναι η μη αυτοματοποιημένη. Πέραν αυτών συζητάμε διαρκώς ε, για την ενεργεία, ειδικότερα μεταξύ των νέων και γνωρίζουμε από την έρευνά μας ε, για τις ευρωπαϊκές δεξιότητες και θέσεις εργασίας ε, ότι δεν απλά δεν υπάρχουν δουλειές, αλλά δεν υπάρχουν καν δουλειέ ποιότητα ή δεξιότητε αχρησιμοποιητέ, τι οποίε μαθαίνει κανεί ε, κατά την εκπαίδευση, αλλά δεν μπορεί να τι εφαρμόσει πουθενά. Από την έρευνά μα, το 25% των εργαζομένων λένε ότι έχουν υπερβολικά πολλά προσόντα και τα 42% των υπαλλήλων δηλώνουν ότι δεν υπάρχει αντιστοίχηση μεταξύ των όσων έμαθαν στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση ε, και των θέσεων εργασία στην αγορά. Και επίσης ξέρουμε ότι από τις θέσεις εργασίας που δεν έχουν καλυφθεί, ξέρουμε ότι για κάθε χίλιους ανέργους στη Γερμανία υπάρχουν τουλάχιστον 400 κενές θέσεις εργασίας, αλλά στην Ελλάδα μόνο 70. Γνωρίζουμε και το γεγονός ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο πολλών ανθρώπων που εγκαταλείπουν πρόωρα τις σπουδέ του. Ε, και επίση ε, έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που δεν βρίσκονται σε φάση εκπαίδευση ή κατάρτιση. Ε, κάτι άλλο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως οργανισμός ε, είναι η εργασιακή φτώχεια, έτσι όπως ονομάζεται, ε, δηλαδή η απουσία θέσεων εργασίας ποιότητας, δηλαδή όταν λέμε ότι δεν αρκεί να έχει κανείς μια δουλειά, αλλά πρέπει η δουλειά αυτή να του παρέχει και μια αξιοπρεπή ζωή. Και το, ο τρίτος παράγοντας είναι η, η κρίση των προσφύγων, όπως ξέρετε είναι απεσιόδοξα τα πράγματα στην Ευρώπη για πολλούς νέους αυτή τη στιγμή αλλά αποτελεί και φάρο ελπίδας για τους μετανάστες που έρχονται εδώ. Οπότε χρειαζόμαστε αλληλεγγύη ε, τόσο για αυτούς που ζουν εδώ όσο και για αυτούς που έρχονται να ζήσουν. Έτσι λοιπόν διαρκώς ε, κάνουμε το δεύτερο ερώτημα. Ποιος είναι ο σκοπός, τι προσφέρει παραπάνω ένας οργανισμός σαν τον ΣΕΔΕΦΟ όσον αναφορά αυτές τις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Αν δείτε το πρόγραμμα εργασιών μας και τα προϊόντα που παρέχουμε μέσα στα ε, έτη, θα δείτε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να οικοδομήσουμε μια ισχυρή κουλτούρα απασχολησιμότητας, μια φιλοσοφία απασχολησιμότητας. Ε, έχουμε στο νου μας τα παραδοτέα της Ρήγα, τα οποία ήταν πέντε ε, και τα οποία ε, συμφώνησαν οι Υπουργοί Παιδείας στη Ρήγα από τώρα μέχρι το 2020, δηλαδή την πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, εργασία ε, βασικές ε, ε, δεξιότητες, εκπαίδευση για διδάσκοντες και μεγαλύτερη ποιότητα στα όσα παρέχουμε στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση. Ο λόγος για τον οποίο προσθέτουμε αξίες είναι για να αναδείξουμε τις δυνατότητες που, που υπάρχουν στην αγορά. Οπότε οι βασικές δεξιότητες ε, σε θέματα πληροφορικής είναι, βασικ... είναι ουσιαστικές για τους νέους. Επίσης προωθούμε διάφορα εργαλεία που διευκολύνουν τη κινητικότητα μεταξύ νέων ε, και εντός των χωρών τους και μεταξύ των χωρών. Και τέλος θέλουμε περισσότερη χρηματοδότηση για τα προγράμματα επαγγελματική κατάρτισης και εκπαίδευση στην Ευρώπη. Όπως γνωρίζετε πολύ, ε, αν δει κανείς το Εράσμος και πώς γίνεται η κατανομή των κονδυλίων, θα δείτε ότι ευνοείται η τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με την επαγγελματική καταρτιστική εκπαίδευση. Ε, με διαφορά 43 και 22% προς ποια κατεύθυνση κινούμαστε τώρα. Κινούμαστε προς την ανάπτυξη περισσότερων ε, θεμελιωδών δεξιοτήτων που θα πρέπει ο κόσμος να έχει όταν παίρνει το πτυχίο του ή το διπλωμά του Επίσης θέλουμε εκπαίδευση για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η διαβίου μάθηση είναι σημαντική, σημαντικός παράγοντας και θέλουμε να προωθήσουμε περισσότερο την εκμάθηση μέσω της πράξης. Οπότε να προωθήσουμε τις πρακτικές ασκήσεις στο πλαίσιο της κατάρτισης. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν στο Διοικητικό μας και εμεί ε, διευθύνουμε τι εργασίε και συνεργαζόμαστε μαζί του για να προωθήσουμε την έρευνα, την ανάλυση και άλλε ειδικευμένε γνώσει και δραστηριότητε που παρέχουν στην Κομισιόν, το Κοινοβούλιο και του Οργανισμού Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδέε και πολιτικές, ε, ε, ιδέες για πολιτικές που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κατάσταση. Το 2015 ήταν ένα ξεχωριστό έτος. Γιορτάσαμε τη 14η μας επέτειο με μια σειρά δραστηριοτήτων μαζί με τις ΕΔΕΦΟΠ και είπα το έτος εκείνο ε, θέλαμε να προωθήσουμε όσο γίνεται το περισσότερο τα συμπεράσματα της ΡΙΓΑ, το αναθεωρημένο εκπαίδευση και ε, κατάρτιση 2020, ένα εργαλείο για να αναβαθμίσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Αυτό σημαίνει ότι ε, εργαζόμαστε υπέρ της βελτιωση της απασχολησιμότητας των νέων. Επίσης, από το 2015 κάναμε μια διοργάνωση των διαφόρων τμήματων μα ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα σε ανάγκε τη Κομισιόν, του Κοινοβουλίου και των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Και σήμερα τα τρία μα τμήματα ανταποκρίνονται στα όσα πρέπει να αλλάξουν ε, στην υποστήριξη τη αποσχολησιμότητας και στη σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των όσων μαθαίνει κανεί στην επίσημη εκπαίδευση και στα σχολεία και των όσων υπάρχουν στην αγορά εργασία και τρίτον η ανάπτυξη δεξιοτήτων εντός της αγοράς. Ε, προσπαθούμε να έχουμε και μια προοπτική, τι εικόνα θα έχει αγορά σε ορισμένα χρόνια από τώρα, ώστε να ανταποκρίνεται αυτά που διδάσκονται στι σχολές ε, στις απαιτήσει της αγοράς εργασίας. Αυτό μεταφράζεται σε νέε δραστηριότητε όπω φόρα χάραξη πολιτική, όπου τα κράτη-μέλη και διάφοροι εταίροι συμμετέχουν. Κάνουμε αναθεωρήσει των πρακτικών ασκήσεων. Πέρσι το κάνουμε με τη Μάλτα και τη Λιθουανία φέτος, ξεκινάμε με την Ελλάδα, τη Σλοβενία και την Ιταλία. Επίση έχουμε δημοσιεύσει, όπω είπα προηγουμένω, την έρευνα ε, θέσεων εργασία και δεξιοτήτων. Έχουμε τη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων για πρακτικέ ασκήσει. Ε, όλα αυτά μας δίνουν μια νέα προοπτική. Πέρυσι είχαμε 49 δημοσιεύματα, 27 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα μας 6.900 ε, άνθρωποι ε, κατέβασαν ε, δημοσιεύματά μας και 4.099 άνθρωποι μας δημοσίευσαν, μας ανέφεραν στα δημοσιεύματά τους. Τώρα θα έχουμε ένα νέο έγγραφο το οποίο θα αναφερθεί στις νέες γνώσεις που χρειαζόμαστε την ανάλυση πολιτικών και την παρακολούθηση των τεκτενόμενων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θέλουμε να δράσουμε ως δημεσολαβητές γνώσεις ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό που παράγουμε εμείς απορροφάται από το σύστημα και δίνει τα σωστά αποτελέσματα. Θα θέλαμε να βοηθήσουμε τους θεσμούς να διαμορφώσουν, να αναβαθμίσουν και να, την, την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση για να δημιουργήσουν ανθρώπους καταλληλότερους για την αγορά ε, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική ένταξη, την ε, αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων, την αντιμετώπιση των πρώιμων αναχωρήσεων από τα σχολεία και την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων. Αυτά είναι τα βασικά προγράμματα που θα προωθήσουμε του χρόνου. Φυσικά βοηθάμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαμορφώσει τη νέα ατζέντα για τις δεξιότητες που θα ξεκινήσει το Μάιο φέτος. Τέλος, ε, όλοι μας ε, λίγο πολύ ζούμε σε έναν κόσμο στατιστικών στοιχείων, εκθέσεων, προβλέψεων, συγκρίσεων και αναλύσεων, αλλά ο κόσμος που βρίσκεται έξω από εδώ ζει σε ένα διαφορετικό κόσμο και από εμά περιμένει να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες του να βρει κανεί δουλειά, να ζει μια αξιοπρεπή ζωή, να διασφαλίσει το μέλλον του. Αυτή είναι η δική μας επιστολή ως ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Αυτή η αναντιστοιχία που βλέπουμε στην κοινωνία είναι αναντιστοιχία μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης και χώρου εργασίας. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε ως οργανισμός για να φέρουμε τους δύο αυτούς κόσμους πλησιέστερα. Από τώρα μέχρι το 2020 βασικός μας σκοπός είναι να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να σκέφτονται ευρωπαϊκά αλλά να δρουν τοπικά, να δρουν ε, ε, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκεί όπου ο κόσμο ε, μαθαίνει και θέλει να συνεχίσει να μαθαίνει και να λαμβάνει δεξιότητες και ικανότητες που θα χρειαστεί στο μέλλον. Μια κινέζικη παροιμία που βρήκα σε κάποιο βιβλίο λέει ότι όταν φυσάει ο άνεμος άλλοι χτίζουν τείχους και άλλοι χτίζουν ανεμόμυλους. Ελπίζω λοιπόν η Σεντεφόπ να παράγει αυτή την ενέργεια για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση. Όπως και Κριστά και εμείς ε, ε, υφιστάμεθα τώρα περικοπές προσωπικού και κονδυλίων και προσπαθούμε να ανακατευθύνουμε τις εργασίες μας ώστε να παράγουμε την ίδια ορμή με αυτή που θέλουμε να παράγουμε. Και ελπίζουμε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και η κατάρτιση για μας και για σας θα αποτελέσει το μήνυμα που θα στείλουμε στους πολίτες μας για να σώσουμε τις ζωές τους και να επενδύσουμε στο μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, James Καγέχα. Και τώρα. Και τώρα αλλάζει το φίλο του μιλητή και είναι Μαντλίν Σέρμπαν. Σας ευχαριστώ όλους για την πρόσκληση αυτή για να σας παρουσιάσω την έκθεση του 15 και μερικές από τις ιδέες μας για το 16. Θέλω να παρουσιάσω το ETF για να σας πω ότι είμαστε ο μόνος φορέας της Ένωσης που χρηματοδοτείται από το κεφάλαιο 4 του προϋπολογισμού. Η Ευρώπη στον κόσμο. Όπως είπε και ο συνάδελφος στο ΣΕΝΤΕΦΟΠ, γιατί χρειάζεται ένας φορέας για να εργάζεται κανείς για το ανθρώπινο δυναμικό στην Ευρώπη. Γιατί χρειάζεται ένας φορέας για το ανθρώπινο δυναμικό σε μια Ευρώπη στον κόσμο. Γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι μόνο η σκληρή δύναμη που είναι αναγκαία στις διεθνείς σχέσεις. Χρειάζεται και η ήπια δύναμη. Και το ανθρώπινο δυναμικό είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στις σχέσεις που έχουμε με πολλές τρίτες χώρες. Όταν λέμε για την Ευρώπη στον κόσμο, το συνδέουμε πάντα με την παγκοσμιοποίηση και πώς μπορεί να συνεισφέρει η Ένωση. Η Ένωση και μέσω και του δικού μας φορέα με την ε, μετριόφρονα συμμετοχή μας ε, είναι να εκπολιτήσουμε την παγκοσμιοποίηση. Όπως είπε και ο Πασκάλ Λαμή που ήταν επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου του πρόεδρου Ντελόρ, ε, η Ευρώπη πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει καλύτερη ισορροπία μεταξύ του κεφαλαίου που είναι στη Δύση, που, συγγνώμη, στην, ε, στον υπόλοιπο κόσμο και στην ελευθερία του συνέρχεστε και συνεταιρίζεστε. Θέλουμε λοιπόν όλες οι χώρες να δώσουν ένα μέλλον για τους πολίτες τους επιτόπου και τονίζω επιτόπου. Η σταθεροποίηση που αναφέρεται σε όλες τις πολιτικές γειτονίες πρέπει να εστιάζεται στη δυνατότητα κάθε χώρας να σταθεροποιηθεί και να δώσει προοπτική στους πολίτες της να ζουν εκεί και πρέπει επίσης να τους δίνει τη δυνατότητα ότι αν κάποιος πολίτης θέλει να μετακινηθεί και πιστεύουμε στην ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών τότε θα πρέπει να υπάρχει μια διαχείριση των νομίμων δυνατοτήτων μετανάστευσης και είναι και αυτό στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας το 2015 συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό που καλούμε το ε, επιχειρηματικό συνεχές στις χώρες αυτές. Τι εννοούμε. Για να μπορέσουν να επιτύχουν σταθεροποίηση οι τρίτες χώρες πρέπει να έχουμε μια πολιτική για την επιχειρηματικότητα, για την ε, ανάληψη κινδύνων, για να μπορεί κανείς να προβλέψει τις επερχόμενες προκλήσεις. Να είναι δηλαδή οι θεσμοί που λειτουργούν στις χώρες να έχουν επιχειρηματικό πνεύμα και να έχουν επίσης την αναγκαία άντοχη για να μπορέσουν να προσαρμοστούν και να βρίσκουν λύσεις. Επίσης οι κοινότητες των χωρών θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσουν, να αξιοποιήσουν το ταλέντο, το δυναμικό, να υπάρχει δυνατότητα καινοτομία για να, εξυπηρετούν, να υπηρετούν τους πολίτες. Και επίσης και οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει να έχουν επιχειρηματικό πνεύμα. Όπως θα είδατε σε αυτή την παρουσίαση τεσσάρων σελίδων των κυριωτέρων επιτευγμάτων του 2015 για την διακυβέρνηση και την εφαρμογή των δημοσίων πολιτικών πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι όσο πιο διαφανής και όσο πιο υπεύθυνη γίνεται. Και όταν λέμε διαφανής, όχι μόνο από οικονομική πλευρά, όλες οι δημοτικές, ε, συγγνώμη, οι δημόσιες πολιτικές πρέπει να έχουν κατεύθυνση προς την δημιουργία αξίας προς όφελος όλης της κοινωνίας. Στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση αναφερόμεθα στην εργασία μας στο Μαρόκο, την Τινησία, σε περιφερειακό επίπεδο. Δηλαδή δεν πάμε μόνο στις πρωτεύουσε, αλλά πολύ κοντά στο νότο της ε, Τινησίας, κοντά στα σύνορα με τη Λιβύη, ούτω ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι θεσμοί που υπάρχουν εκεί έχουν δυνατότητα να πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους, μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους για να συντονίσουν τις προσπάθειες, προσπάθειες τους. Το κάναμε στο Μεντίν και στο Γκαμπές. Και ως συνέχιση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει άλλες 8 περιφέρειες από εφέτος. Δεν εγκαταλείπουμε την βοήθεια πολιτικής ε, σε κεντρικό επίπεδο, αλλά θέλουμε οι εξελίξεις αυτές να γίνονται και σε τοπικό επίπεδο σε μικρότερο βαθμό είμαστε παρόντες και στην Αλγερία όπου οι επιχειρηματίες έλαβαν στήριξη και μπορούν να προσφέρουν εναλλακτικέ λύσεις ε, στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Την ανάγκη δηλαδή διαφοροποίησης ε, της οικονομίας τους που βασίζεται πολύ στην οικονομία, στην, ε, συγγνώμη, στο πετρέλαιο. Και επειδή έχει μειωθεί πολύ η τιμή του πετρελαίου, χρειάζονται εναλλακτικές οικονομικές δυνατότητες για να υπάρξει εισόδημα για τους πολίτες σε σχέση με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Να αναφέρω μια προτεραιότητα που ελπίζω και εσείς να τη βρείτε χρήσιμη. Στήριξη των χωρών του Μαγκρέμπ, Μαρόκο, Τινησία και Αλγερία. Οι χώρες αυτές θέλουν να συνεργαστούν με, τους, ε, με τον ιδιωτικό τομέα στις χώρες τους, αλλά και με την ευρωπαϊκή βιομηχανία, την ευρωπαϊκή οικονομία που επενδύει στις χώρες τους ούτως ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους εργαζόμενοι. Έχει αναφερθεί αυτό. Αλλά εάν οι χώρες αυτές θέλουν να βρουν ευκαιρίες, δυστυχώς δεν υπάρχουν πόροι για να τους δώσουν ευκαιρίες. Ίσως με τη δική σας στήριξη ως Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσουμε το μέσο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας ούτως ώστε να υπάρξουν δυνατότητες ε, να εκπαιδευτούν σε ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις ή σε ε, τοπικές επιχειρήσεις. Έχουμε λοιπόν μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση με οριζόντια βάση. Κάνουμε πολλά για να αναπτύξουμε τις δυνατότητες κεντρικής Ασίας. Εκεί προσπαθούμε να αναπτύξουμε την εκπαίδευση. Οι χώρες αυτές, ξέρετε, είναι πολύ συγκεντρωτικές της κεντρικής Ασίας. Αλλά εδώ και μερικά χρόνια προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε την εκπαίδευση, να χτίσουμε σχολεία μέσω μιας διακυβέρνησης που να συμμετέχουν και οι τοπικοί φορείς να υπάρχει επαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση για τους νέους. Άλλες θα πάνε καλύτερα από άλλες. Θέλουμε όμως να τους δώσουμε ευκαιρία να μάθουν και από τους ε, ας πούμε τους εργαζόμενους με περισσότερη πείρα. Έχουμε λοιπόν μια πλατφόρμα για την Κεντρική Ασία. Στηρίζουμε έτσι την ενωσιακή ατζέντα, το ενωσιακό θεματολόγιο. Για την Ανατολική Ευρώπη θα αναφερθώ στην εργασία που κάναμε για να προσαρμοστούν οι δεξιότητες στη ζήτηση. Στην περίπτωση της Ουκρανίας για παράδειγμα. Οι εργοδότες όντως έχουν αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες, έχουν καταφέρει να συνεργαστούν για να εντοπίσουν τις ε, ανάγκες τους και χαίρομαι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι από την Ουκρανία παρόντες και αυτό που κάνει για να αναπτύξει νέες δεξιότητες η Ουκρανία είναι πραγματικά αξιόλογο αλλά και άλλες χώρες στην περιοχή η Γεωργία για παράδειγμα η Μολδαβία μαθαίνουν πώς να ξεκινήσει ο κοινωνικός διάλογος για να προωθήσουν την επαγγελματική κατάρτιση. Αλλά πρέπει επίσης να τονίσω ότι η Γεωργία ε, έχει την καλύτερη δημόσια δίκηση στην περιοχή. Γι' αυτό στηρίζουμε τη χώρα για να διασφαλίσουμε την συμμετοχή ευρυτέρων στρωμάτων στην επαγγελματική κατάρτιση και η χώρα αυτή είχε εξαιρετικά αποτελέσματα στη χορήγηση ευκαιριών στα άτομα με ειδικέ ανάγκες για να έχουν πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση. Ίσως να είναι συνηθισμένο αυτό στην Ευρώπη, αλλά σε πολλές άλλες χώρες δεν είναι. Δεν έχουν όλοι πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου εκπαίδευση. Δεν υπάρχει ισότητα και ισότητα ευκαιριών. Για τη Μονταβία έχουμε ένα παρατηρητήριο για την αγορά εργασίας γιατί η χώρα αυτή έχει ανάγκη μεγάλων διαθρωτικών αλλαγών. Θέλουμε να τη βοηθήσουμε να μπορέσει να εργαστεί σε τοπικό επίπεδο, καθώς και σε κλαδικό. Για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία. Έχουμε κάνει πολλά μέσω της νομοθετικής πράξης για την αποτίμηση της ε, εργασίας των μικρών επιχειρήσεων. Η οργάνωσή μας, η TF, εδώ και χρόνια έχει αναλάβει την ευθύνη να αποτιμά την εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα και την ε, απόκτηση δεξιοτήτων σε όλες τις περιοχές εκτός από την Κεντρική Ασία. Και τώρα ασχολούμεθα με τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία. Κάνουμε έκθεση για αυτή την περιοχή. Αυτά που σας λέω βεβαίως είναι γνωστά, δεν υπάρχει θέμα εμπιστευτικότητας. Θέλω λοιπόν να σε ενημερώσω ότι δυστυχώς παρατηρούμε ότι δεν δημιουργούνται πάρα πολύ λίγες θέσεις εργασίας από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν φέτος θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης για να δούμε πώς θα στηρίξουμε καλύτερα τον ιδιωτικό τομέα για να υπάρξουν αποτελέσματα. Επίσης, ε, το ευρωπαϊκό μέσο που αξιοποιούν τα κράτη-μέλη για την εγγύηση της, ε, των θέσεων απασχόληση για την νεότητα, που αξιοποιείται και στην Τουρκία, επηρεάζει επίσης τις δραστηριότητες στα Δυτικά Βαλκάνια. Το 2016 θα συνεχίσουμε λοιπόν να εργαζόμεθα σε τοπικό επίπεδο για να αποκτήσουν δεξιότητες και προσόντα οι εργαζόμενοι και για να εκπαιδευτούν στην επιχειρηματικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Επιτροπή σας για τη στήριξή της ε, το, ε, το περασμένο έτος, για την εργασία που κάναμε για τη μετανάστευση και που παρουσιάσαμε σε προηγούμενες συνεδριάσεις. Και σας ευχαριστώ και για την εργασία που παρουσιάσαμε μαζί με τον εκπρόσωπό σας στο Τωρίνο για την αποτίμηση των δημοσίων πολιτικών. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρό σας που μας προσκάλεσε να συμβάλλουμε σε αυτή τη συζήτηση για, τα για τα, αυτά που κάνουμε στα διάφορα κράτη-μέλη και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό και προσφυγικό περισσότερο. Και ευχαριστώ τον παρατηρητή σας στο ε, διοικητικό μας συμβούλιο, την κυρία Edith Bauer. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε τρεις ανεξάρτητους ε, οι δήμονες που συμμετέχουν στο Διοικητικό μας Συμβούλιο. Και ξέρω ότι θα έρθετε να μας επισκεφτείτε και ελπίζω λοιπόν να έρθετε και ελπίζουμε να σας δούμε όλους για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να, να αλλάξουμε όχι μόνο την Ευρώπη αλλά συνολικότερα τον πλανήτη. Ευχαριστώ Μάντλιν Σέρμπαν. Ο κύριος Χουάν Μενίντες Βαλδές έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι άλλη μια χρονιά εδώ μαζί σας με τους επικεφαλείς των τριών άλλων οργανισμών και να σας παρουσιάσω τα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Τρίματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας το 2015 και θα σας πω τι σχεδιάζουμε να κάνουμε το 2016. Γνωρίζετε ποιο είναι ο ρόλος της Eurofound. Είμαστε περίπου 108 άτομα ε, κυρίως ε, στο Δουβλίνο με ένα μικρό γραφείο στις Βρυξέλλες με προϋπολογισμό 20 εκατομμυρίων με στόχο να ε, προσφέρουμε γνώσεις όσον αφορά την ανάπτυξη πολιτικών για την εργασία και τις κοινωνικές πολιτικές. Τέσσερα στοιχεία για πέρσι και φέτος θα ήθελα να αναφέρω. Ε, μαζί με το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, όπως και το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, ε, ε, και εμείς πέρσι γιορτάσαμε την 30η επέτειο της παρουσίας μας. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για να ξανασκεφτούμε πώς θα μπορούσαμε να επιτυχάνουμε το, τους στόχους μας. Επίσης συμμετείχαμε στο δίκτυο Ευρωπαϊκών Οργανισμών που πλέον συμπεριλαμβάνει 44 οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς προτείναμε την έγκριση της ε, στρατηγικής ατζέντα. Αν θέλετε μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, ε, για πρώτη φορά ε, παρουσιάσαμε το νέο εναρμονισμένο πρότυπο για τον προγραμματισμό μας για την περίοδο έως το 2020 και έτσι παρουσιάσαμε λοιπόν το έργο μας για το 2016, για το 2017 έως και το 2020 και το 2016 θα δείτε πιθανότατα μια πρόταση της Κομισιόν για την ε, προσαρμογή του κανονισμού ε, με βάση την ε, συμφωνία που επιτεύχθη μεταξύ των αποκεντρωμένων οργανισμών. Οι δραστηριότητε της Eurofound που είναι οι πιο γνωστές είναι οι τρεις ε, πανευρωπαϊκές μελέτες που διεξάγουμε. Φέτος θα ξεκινήσουμε το επιτόπιο έργο στο τέλος της, ε, της φετινής χρονιάς για την μελέτη για την ε, ποιότητα της ζωής. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί η παρουσίαση των πορισμάτων θα γίνει από του χρόνου και τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ε, την μελέτη για τις συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη. Πέρσι ε, διεξέγαμε την έκτη έρευνα, ε, σχετική έρευνα για την παρακολούθηση των συνθήκων εργασίας στην Ευρώπη, κάτι που έχει ξεκινήσει από το 1990 και εμείς καταλήξαμε σε συγκεκριμένα πορίσματα για τις τάσεις στην Ευρώπη και αυτό τον καιρό ε, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε και ελπίζουμε τον Νοέμβριο φέτος να καταφέρουμε να σας παρουσιάσουμε και εδώ στο Κοινοβούλιο την ανάλυση μας για τα συνολικά στοιχεία. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η μελέτη για τις συνθήκες εργασίας ε, βασίζεται σε πληροφορίες όχι μόνο από, τις ευρωπαϊκές, από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλά και από τον ε, ΟΑΣΑ και προσπαθούμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με τον ILO και άλλα ερευνητικά κέντρα για να καλύπτουμε την Κίνα και τις ΗΠΑ, άλλες χώρες δηλαδή, για να μπορέσουμε το 2017 να υποβάλουμε και μια παγκόσμια έκθεση. Πέρσι συλλέξαμε ε, λεπτομερέστερες πληροφορίες για τις πραγματικότητες που ε, βρίσκονται πίσω από την περίπλοκη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ε, αυτοαπασχολούμενοι και φέτος θα υποβάλουμε έκθεση για τις διάφορες καταστάσεις που ε, επικρατούν στον τομέα των ε, αυτοαπασχολουμένων. Επίσης θα εξετάσουμε τα ζητήματα που σχετίζονται με τον χρόνο εργασίας, με το θόλωμα των γραμμών και των ορίων μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματική ζωής θα υπάρξει και διαβούλευση ε, με την Κομισιόν και κάτι που αναφέραμε εμείς ήδη στο Κοινοβούλιο πέρσι με την... αφορούσε την ε, άδεια μητρότητας και πατρότητας. Έχουμε και καλά νέα. Τα περισσότερα κράτη-μέλη ε, δίνουν περισσότερη άδεια ε, από την υποχρεωτική περίοδο των ε, δύο εβδομάδων, αλλά υπάρχουν ακόμα δύο κράτη-μέλη που δεν έχουν υποχρεωτική άδεια μητρότητας και πατρότητας. Ο χρόνος εργασίας είναι ένα σημαντικό θέμα όπου τα όρια θολώνουν και εμείς με το μηχανισμό παρακολούθησης ε, παρακολουθούμε πολύ στενά τις, αγοράς, τις αγορές εργασίας. Εξετάζουμε και διάφορες νέες μορφές εργασίας, ε, νέες μορφές εργασίας, γιατί έχει αλλάξει η σχέση ένα προς ένα μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου και προσαρμόζονται και εμφανίζονται νέες πραγματικότητες ε, και ε, αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται βεβαίως και στις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά εμείς παίρνουμε υπόψη και τα τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης ε, στο πλαίσιο ενός ποιητικού προγράμματος που μας ανέθεσε το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν ε, με αντικείμενο το μέλλον της μεταποίησης και της απασχόλησης στον τομέα και την ε, κατάσταση σε περιφερειακό επίπεδο. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις διαστρωτικές αλλαγές που συνεχίζουν να συμβαίνουν στην αγορά εργασίας μέσα από τα μόνιμα εργαλεία μας, αλλά φέτος επίσης θα κάνουμε και μια σε βάθος ανάλυση των ε, αποθεμάτων των ε, ε, αγορών εργασίας, όχι μόνο των ανέργων και των μακροχρόνια ανέργων, αλλά και εκείνων που είναι ανενεργοί. Επίσης εξετάζουμε τις πολιτικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για να επανέλθουν οι άνθρωποι αυτοί στην, ε, στην εργασία. Και βασιζόμενοι στο, στο ε, έργο του παρελθόντος που έχουμε κάνει, εξετάζοντας τους νέους ανθρώπους, θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε και το ζήτημα της μακροχρόνιας ανεργίας των νέων. Ε, η μετανάστευση είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα το τελευταίο διάστημα και εμείς έχουμε δημοσιεύσει μια σχετική έρευνα Όσον αφορά τον ε, αντίκτυπο ε, που έχουν ε, οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι από τις χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης σε άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν πλήττουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας των άλλων κρατών. Συνολικά πολίτες ε, αυτών των νέων χωρών μετά την διεύρυνση συμβάλλουν θετικά στο ισοζύγιο για τα κοινωνικά συστήματα ε, προστασίας και φέτος θα αναλύσουμε την κατάσταση των ε, μετακινούμενων και των μεταναστών εργατών και για την ένταξη των ε, μεταναστών, προσφύγων και ετούντων έσυλο έπειτα από αίτημα του Διευθυντικού μας Συμβουλίου. Μια τρίτη μελέτη που κάναμε αφορά την, ε, τις ε, ευρωπαϊκές εταιρείες και φέτος επικεντρωθήκαμε σε συγκεκριμένα στοιχεία και αυτό που θέλω να σας επισημάνω είναι ότι βρισκόμαστε σε συζητήσεις με το ΣΕΝΤΕΦΟΠ αυτό το διάστημα να εξετάσουμε μήπως θα μπορούσαμε από κοινού να διοργανώσουμε την νέα ε, ευρωπαϊκή έρευνα για τις εταιρείε. Νομίζω ότι ε, αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να καταλήξουμε σε χρήσιμα και θετικά αποτελέσματα αλλά και να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους οι οργανισμοί. Στην έρευνα αυτή για τις ευρωπαϊκές εταιρείες κοιτάζουμε και τις συμμετοχές, τη συμμετοχή των εταιρεών στον κοινωνικό ε, διάλογο και η Κομισιόν έχει καταβάλει συγκεκριμένε προσπάθειες προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία αυτός ο κοινωνικός διάλογος. Ε, συγκεκριμένο θέμα που έχει δημοσιευθεί ε, και το οποίο έχουμε εξετάσει εμείς είναι και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η εικόνα ε, είναι διαφορετική από κράτος μέλος σε κράτος ε, μέλος. Υπάρχει μόνο ένα κράτος μέλος το οποίο η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική. Παρ' όλα αυτά γίνονται πρόοδοι και η Κομισιόν καταβάλει προσπάθειες. Επίσης, ε, υπάρχει ο διακλαδικός ε, διάλογος ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εμείς βελτιώνουμε και τις διαβάσεις δεδομένου μας για τις βιομηχανικές σχέσεις. Να σας πω και τι θα γίνει το 2017 με 2020. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στους τέσσερις τομείς που ε, είναι στην αρμοδιότητά μας, αλλά θα εξετάσουμε και τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στον κόσμο της εργασίας και της απασχόλησης και θα παρακολουθήσουμε την σύγκληση ή την απόκληση όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, εργασίας στην Ευρώπη ε, υπό το φως και των ε, εξελίξεων των τελευταίων χρόνων. Να σας πω και κάποια στοιχεία. Το 99,9% του προϋπολογισμού μας ε, αξιοποιήθηκε πέρσι, 229 δημοσιεύσεις, 129 δημοσιεύσεις, 300 20 ε, ε, έγγραφα πολιτικής, 59 ε, από αυτό το κοινοβούλιο και πάνω από χίλιες εκθέσεις που ελήφθησαν από την ιστοσελίδα μας. Και τέλος, να σας πω και εγώ για τους πόρους του, του οργανισμού μας. Ήδη εμείς έχουμε περικόψει κατά 5% το προσωπικό μας, το ίδιο σχήκε και για τους άλλους οργανισμούς. Έχουμε ήδη ε, μειώσει κατά 6% το προσωπικό φέτος και το 10% που ε, μας έχει ζητηθεί θα εφαρμοστεί πριν από το 2018 αλλά ας μην έχουμε υπερβολικές ε, προσδοκίες και ας μην θεωρούμε ότι αυτό θα ε, έχει ουδέτερο αντίκτυπο. Φυσικά και θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις αυτής της μείωσης. Υπάρχουν ήδη κάποιες συζητήσεις στα, στις ομάδες εργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Η επόμενη θα γίνει 13 Μαρτίου που αφορά την αύξηση της αποδοτικότητας, την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων, ε, όπου και το Κοινοβούλιο ε, θα μπορέσει να τοποθετηθεί αν ε, οι πολιτικές απασχόλησης θα έχουν την ίδια ή υψηλότερη ή χαμηλότερη προτεραιότητα σε σχέση με, παλιό, με παλιά. Και εδώ οι, οργανισμού, οι οργανισμοί πιστεύω ότι θα πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε δεσμευμένοι και αφοσιωμένοι στο να επιτύχουμε τους στόχους μας και να καταδείξουμε ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με βάση τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ και με αυτό ε, τελειώσαμε με τις παρουσιάσεις των τεσσάρων οργανισμών. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Ο David Κάς έχει το λόγο. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Να σας ευχαριστήσω επίσης και για το έργο σας, για την εκκρίσιμη σημασία ιδιαίτερα χρήσιμα εργαλεία για τις καθημερινές μας εργασίες. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά τους νέους. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι νέοι έχουν πλέον πολλούς τρόπους για να μάθουν πράγματα εξωσχολικά. Ενδιαφέρον θα ήταν να δούμε κατά πόσο έχουν γίνει μελέτες ή έρευνες όσον αφορά πρακτικές ασκήσεις, προγράμματα μαθητείας και πώς αυτά ωφελούν τις επιχειρήσεις. Ε, ε, αν όχι υπάρχει σχέδιο να πραγματοποιηθεί κάποια μελέτη και να ενθαρρυνθούν οι εταιρείε να βοηθούν του νέου να αποκτούν νέε επαγγελματικέ εμπειρίε. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι προς τον κύριο James Καλιαχά τη ΣΕΔΕΦΟ που μίλησε για τους μετανάστες και του πρόσφυγες και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα. Η επικύρωση άτυπης και μη τυπικής εκμάθησης ε, είναι μια πρόκληση σε όλα τα επίπεδα αλλά πιστεύω θα δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο όσο, όταν αφορά τους πρόσφυγες που φτάνουν στις ακτές μας. Υπάρχει κάποια μελέτη της ΕΔΕΦΟΠ για το πώς θα γίνει η επικύρωση ε, και άλλες πολιτικές επαγγελματικές και ε, ε κατάρτισης και εκπαίδευσης για τους πρόσφυγες και η τρίτη μου ερώτηση η ΣΕΔΕΦΟΠ ε, εργάζεται σε κανένα πρόγραμμα για την κατάρτιση και την ένταξη των προσφύγων πιο συγκεκριμένα έχει γίνει κάποια ανάλυση, κάποια μελέτη για το είδος της ε, εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα χρειαστούν ενδεχομένω οι πρόσφυγες για να ενταχθούν πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ιούτα Στάινροκ. Καταρχάς ε, ευχαριστώ όλους τους φορείς και παρακαλώ να δώσετε τα ευχαριστήριά μας, να εκφράσετε την ευγνωμοσύνη μας και προς τους συνεργάτες σας Όλοι όσοι έρχονται κάθε χρονιά σε αυτή τη συνάντηση ξέρουν πόσο μας, βοηθεί, πόσο μας βοηθάει αυτή η εργασία που κάνουν αυτοί οι θεσμοί. Οι συνάδελφοι εδώ ίσως να μην ξέρουν πολύ καλά την εργασία αυτών των φορέων, αλλά εγώ και η ομάδα μου ασχολούνται πάρα πολύ με τις μελέτες, με την πληροφόρηση που λαμβάνουμε, με τις δραστηριότητες τους, είναι απαραίτητες. Ε, πιστεύω ότι εκπληρώνετε τα καθήκοντά σας με πολύ καλό τρόπο. Ε, πάντα συζητάμε για νέα καθήκοντα για όλους αυτούς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Θα είχε επιπτώσεις και σε εσά εάν είχατε και εσείς ε, διεύρυνση των αρμοδιοτήτων σας. Να σχολιάσω τώρα. Η εκπαίδευση και εκδημοκρατισμό στις υποψήφιες χώρες και τρίτες χώρες. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά. Όποιος παρακολουθεί τα νέα. Θα ήθελα να μου πείτε πού υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη για δράση, γιατί υποθέτω ότι δεν έχετε απεριόριστα μέσα, απεριόριστους πόρους για να λύσετε όλα τα προβλήματα. Πήγα πρόσφατα και στο Σεντεφόπ στη Θεσσαλονίκη και διαπιστώσαμε ότι το ΣΕΝΤΕΦΟΠ στον τομέα της κατάρτισης, της διαβίου κατάρτισης, της ένταξης των προσφύγων στην αγορά εργασίας αλλά και για την ψηφιοποίηση αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Συμφωνώ με την ερώτηση του συναδέλφου Κάζα, η ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας Μπορείτε να βοηθήσετε τα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό. Να αποκτήσουν δηλαδή ε, τις ιδιότητες, να μπορούν να δίνουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Πρέπει μαζί να κάνουμε κάτι για τον όσα. Πώς αξιοποιούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτά που κάνετε. Συζητάμε για το refit και λέμε πάντα ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ε, υπερβολική γραφειοκρατία. Μήπως θα έπρεπε να καταργήσουμε κάποια νομοθετήματα για να τις υποστηρίξουμε καλύτερα. Ούτως ώστε να έχει και καλύτερη εντύπωση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης για το Eurofound έχει αλλάξει η φύση της εργασίας. Θέλω να μας πείτε πώς την έχετε διαπιστώσει. Συζητάμε τις τελευταίες ε, ε, μέρες εδώ την ε, κινητικότητα εντός της Ένωσης και τα επιδόματα που πρέπει να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι όταν μετακινούνται. Πώς βλέπετε να είναι η κατάσταση. Γιατί έχει να κάνει και με την συζήτηση που είναι τόσο επίκαιρη. Ευχαριστώ και με συγχωρείτε αν μακρηγόρησα. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Η κυρία Μάκιντάρ δεν είναι παρούσα, ούτε η Μαρία Χάρκιν Ρένα Ρόνια Κάρι Α, η Ρένα Τεβίμπα. Για το ECR. Α, για, το, για την Άλτε. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας. Πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις τους. Πολύ ενδιαφέρουσα η ενημέρωση που λάβαμε για την εργασία των οργανισμών αυτών τα τελευταία χρόνια. Να πω τα Αναμφίβολα η κοινωνική Ευρώπη είναι μια έννοια που μας απασχολεί εδώ και καιρό. Ωστόσο, η Ευρώπη δεν πρέπει να χάσει την ανταγωνιστικότητά της ε, σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε συγκεκριμένες δεξιότητες Χρειάζεται να μην υστερούμε άλλων χωρών. Αλλά δυστυχώς υστερούμε από ορισμένε απόψεις. Παράλληλα βέβαια, μας ανησυχεί ιδιαίτερα αυτή η νέα ασθένεια του σημερινού κόσμου το στρες και η ψυχοκοινωνική κίνδυνη στην εργασία αλλά το στρες οφείλεται επίσης στο ότι ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πολύ διαφορετικός από τον κόσμο πριν από 100 χρόνια. Για παράδειγμα, η κυκλοφορία για να πας τη δουλειά σου και να γυρίσεις σπίτι σου, αυτό δημιουργεί τρομερό στρες. Όπως είπε ο κύριος Καγέχα, 42% του πληθυσμού θεωρούν ότι δεν ε, αξιοποιούν τις δεξιότητες ε, που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της σχολικής τους εκπαίδευσης. Δηλαδή ξεκινάς να δουλεύεις και σε αγχώνει το ότι δεν μπορείς να αξιοποιήσεις τα προσόντα σου. Και το 25% που θεωρούν ότι έχουν πολύ ψηλότερα προσόντα από αυτά που απαιτούνται για τη δουλειά τους. Και αυτοί βεβαίως ε, αγχώνονται για αυτό το λόγο. Μία ερώτηση για την κυρία Σλέντλατσεκ. Στις έρευνες που κάνετε, Λάβατε υπόψη και αυτούς τους άλλους παράγοντες βέβαια. Άγχος στην εργασία. Ακούγεται λίγο ε, στενή αντιμετώπιση. Πώς αντιμετωπίσατε τους άλλους παράγοντες άγχους. Και κάτι άλλο για όλους τους προσκεκλημένους μας. Έχετε κάνει μια συνολική μελέτη που να καλύπτει τους τομείς ε, αρμοδιότητας όλων των οργανισμών αυτών για να λάβετε μια συνολικότερη εικόνα. Γιατί από την παρουσίαση του καθενός σας έχω την εντύπωση ότι έχετε κάνει μελέτες που εξετάζουν ε, επιμέρους θέματα. Ποιος θα συνθέτει όλα αυτά σε έναν καμβά. Ευχαριστώ πολύ. Τζίν Ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω και τους προσκεκλημένους για τις εκθέσεις και που μας παρουσίασαν μόλι. Έχω ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα για την Eurofund. Ευχαριστούμε πολύ για το έργο που έχετε επιτελέσει εξετάζοντας όλα τα ζητήματα της κινητικότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ευρήματα που προέκυψαν, τα οποία θα αποδειχθούν πολύ χρήσιμα όσον αφορά τη δεσμή μέτρων για την κινητικότητα των εργαζομένων και κάποια πράγματα που θεωρούμε δεδομένα σε ε, πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Δεύτερον, ε, πολλοί ρώτησαν για το ζήτημα των προσφύγων που θα το αφήσω στην άκρη. Θέλω να ρωτήσω για τις ανάγκες για τους, ε, συγγνώμη, για τους ανθρώπους εκτός εκπαίδευσης, ε, απασχόλησης ή κατάρτισης τους NET. Ε, Έχουμε κάνει εμεί κάποια έρευνα για την Τουρκία. Ξέρω ότι η Eurofund έχει κάνει σχετική έρευνα στο παρελθόν. Είμαι βέβαιο ότι και άλλοι το ερευνούν αυτή τη στιγμή. Πιστεύετε ότι σημειώνεται κάποια βελτίωση ότι μειώνεται ο αριθμός, ότι βελτιώνονται εκεί οι δεξιότητες και οι ευκαιρίες. Ειδικότερα και μάλιστα βάσει των όσων είπε μόλις η συνάδελφος Μρενάτα αν έχουμε αυτό το κενό στην αγορά εργασίας που ακούμε και υπάρχει ο κόσμος ο οποίος εκπαιδεύεται για κάτι και τελικά αυτά που μαθαίνει δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, τι μπορούμε να κάνουμε είτε αυτό είναι αξιολόγηση της αγοράς εργασίας, είτε είναι πρόβλεψη του μέλλοντος της αγοράς εργασίας, ώστε να μπορέσουμε να ε, γεφυρώσουμε αυτά τα χάσματα, διότι ξέρετε... Στα ταξίδια που κάνουμε συναντάμε πολλούς ανθρώπους που συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα κατάρτισης και ο ένας μου λέει ναι ακολουθώ αυτό αλλά δεν εξακολουθώ να μην έχω δουλειά. Κάνουμε κάτι γι' αυτό. Από ό,τι φαίνεται όχι αρκετά. Ε, εσείς λοιπόν θεωρείτε ότι ε, σας ε, ακολουθούν οι εργοδότες. Ε, Εκπαιδεύετε σωστά τον κόσμο για να τους ικανοποιήσετε, για να καλύψετε τις ανάγκες που θα έχουν στις επιχειρήσεις τους. Ευχαριστώ. Για το ENF, Ντομινίκ Μαρτάου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους διαφορετικούς διευθυντές που ήθελαν να μας παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη ερώτηση. Ευχαριστώ. Η Αλεσάνδρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για όλες τις πληροφορίες που ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες όπως και η παρουσίαση. Εγώ θέλω να επιμείνω σε δύο σημεία. Πρώτον, ε, η ε, εκμάθηση, μιλήσετε για την εκμάθηση και θέλω να τονίσω ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί αυτή η εκμάθηση, η μαθητεία, αλλά και να αναπτυχθεί και η κινητικότητα των μαθητευομένων. Σήμερα έχουμε στη διαθέση μας εργαλεία, ειδικότερα το Erasmus Plus, που έχει ως στόχο να ευνοεί τους νέους μαθητευομένους νομίζω και ο διευθυντής του ΣΕΔΕΦΟΠ μίλησε για το Erasmus Plus αλλά όπως γνωρίζουμε όλοι αυτοί οι νέοι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν προσκόμματα που δεν γνωρίζουν άλλες κατηγορίες όπως οι φοιτητές. Εμείς έχουμε δει τα προβλήματα κινητικότητας, τα προβλήματα στέγασης και όλα αυτά σχετίζονται και με το γεγονός ότι οι μαθητευόμενοι είναι συνήθως νεότεροι σε ηλικία από τους φοιτητέ. Οπότε υπάρχει και ένα πρόβλημα του καθεστώτος των μαθητευομένων. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν στις μελέτες σας έχετε εντοπίσει ε, επιπλέον προσκόμματα και αν έχετε βρει πιθανές οδούς ε, ε, επίλυση αυτών των θεμάτων που θα μπορούσατε να μας αναφέρετε. Το δεύτερο στο οποίο θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση είναι οι ικανότητες οι αρμοδιότητες, συγγνώμη, σε διάφορους οργανισμούς στο ΣΕΝΤΕΦΟΠ ε, ε, κάνετε κάποιες μελέτες ε, προοπτικών. Εγώ συχνά πηγαίνω και συναντώ νέου και όταν του λέω ότι ασχολούμαι με ζητήματα απασχόληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μου λένε σε ποιον τομέα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε σήμερα. Εσείς λοιπόν που κάνετε μελέτες, έχετε να απαντήσετε στο ποιες είναι οι ικανότητες που θα εντοπίσουμε σήμερα και οι οποίες θα είναι απαραίτητες αύριο στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Elizabeth Μανοσάτιε επανήλθε οπότε έχει και το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη που βγήκα. Είχα μια ομάδα εκπροσώπων ε, της βιομηχανίας που χάρηκαν ιδιαίτερα που βρέθηκαν εδώ και άκουσαν τις παρουσίες αυτές. Ε, να σας ευχαριστήσω όλους. Εγώ θα συνεχίσω αυτά που μόλις είπε η Αν Σαντέρ. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε να επιλύσουμε σήμερα σε θέμα κατάρτισης είναι το θέμα της οικοδόμησης μεταβιβάσιμων ικανοτήτων Δηλαδή πρέπει να δούμε προς ποιου τομεί πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους νέους ώστε να μπορέσουν να μπουν στην αγορά εργασίας. Εγώ επιπλέον θα... σας παρακαλούσα να μας διαφωτίσετε για τα βασικά κατόφλια ικανοτήτων που είναι απαραίτητα ώστε να μπορεί ένας νέος να μπει στο χώρο στην αγορά εργασίας. Εγκαταλείπω τους συγκεκριμένους τομείς τώρα ε, και αυτή την προβληματική και μετά τις επιμέρους ικανότητες που χρειάζεται να έχει κανείς, κανείς νέος, ώστε να μπορεί να εκμεταλλευτεί την κινητικότητα, τη δυνατότητα κινητικότητας εντός της αγοράς εργασίας. Δηλαδή το να μπει με ε, εφαρμόσιμες ικανότητες στην αγορά εργασίας και να έχει τη δυνατότητα κινητικότητας. Αυτά είναι τα προβλήματα που πρέπει να υπερπηδήσουμε. Ουσιαστικά το πώς περνάει κανείς από μια ε, θεωρητική εκπαίδευση σε μια εκπαίδευση βάση ικανοτήτων. Το δεύτερο, βλέπουμε ότι επικεντρωνόμαστε ε, σε αυτές τις ιδέες των ικανοτήτων και θέλουμε να δούμε πώς ε, θα έχουμε και ατομική εκπαίδευση πέραν των όσων είπαμε. Σε αυτό το τομέα που παρουσιάζονται τόσες λήψεις πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε διότι ξέρουμε ότι σε όλα τα συστήματα παιδείας ε, στην Ευρώπη δημιουργούμε μάζες ανθρώπων και όχι άτομα. Και αυτή η έλλειψη ατόμων οδηγεί στο να έχουμε ανθρώπους ενινητή και ε, ελλείψεις ε, ικανοτήτων. Ευχαριστούμε. Η Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ να ευχαριστώ, σας ευχαριστήσω όλους για τις παρουσιάσεις σας που όντως, όντως ε, μας διευκολύνουν για την εργασία μας. Έχω συγκεκριμένε ερωτήσεις. Κυρία Σεντλάτσεκ, αναφέρατε ότι είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους να φτάσουν μέχρι την ηλικία συνταξιοδότηση σε καλή υγεία, σε καλή κατάσταση. Τι νομίζουν οι εργοδότες. Εμείς μπορούμε να προτείνουμε προγράμματα, αλλά δεν το καταλαβαίνουν αυτό οι εργοδότες ότι πρέπει να συμμετάσχουν στην, ε, στον καθορισμό αυτών των λύσεων δεν θα επιτύχουν αποτελέσματα. Και αυτοί οι γυρεότεροι εργαζόμενοι βεβαίω είναι έμπειροι αλλά δεν είναι πάντα τόσο υγιείς όσο θα ήθελαν ενδεχομένω οι εργοδότες τους. Κύριε Καγέχα, αναφερθήκατε σε προγράμματα κατάρτισης και στην διαβίου μάθηση. Βεβαίω, Εγώ θα ήθελα περισσότερο να χρησιμοποιούμε τον όρο διαβίου ε, εξέλιξης στη σταδιοδρομία. Γιατί ορισμένοι δεν ε, θέλουν τόσο πολύ να τους λέμε ότι πρέπει να μάθουν κι άλλα σε όλη τη διάρκεια της ε, εργασιακής του ζωής. Αλλά βέβαια οπωσδήποτε για να παραμείνεις στην αγορά εργασίας πρέπει σε όλη σου τη ζωή να αναπτύσσεις καινούριε δεξιότητες, να μαθαίνεις περισσότερο. Εκπαιδεύετε λοιπόν και τους επιχειρηματίες. Τους παρέχετε κατάρτιση γιατί πρέπει να μάθουν πώς να διαχειρίζονται σωστά την επιχείρησή τους και πώς να επικοινωνούν σωστά με τους ε, εργαζόμενούς τους. Νομίζω λοιπόν ότι αν ο στόχος ε, της επιχείρησης είναι να πείσει και τους εργαζόμενους ότι πρέπει να συμμερίζονται τους στόχους της επιχείρησης, τότε θα επιτύχει. Τους παρέχεται τέτοια εκπαίδευση. Κυρία Έρμπαν, νομίζω ότι η παρουσίασή σας ήταν αυτή που με ενθουσίασε περισσότερο. Γιατί είπατε ότι πρέπει να διδάξουμε την επιχειρηματικότητα. Πιστεύω ότι η καταπολέμηση της φτώχειας και της ε, ανεργίας μπορεί να γίνει μόνο μέσω της εκμάθησης επιχειρηματικού πνεύματος, ιδίως βέβαια στους νέους. Προσπαθείτε λοιπόν να αλλάξουν ε, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ούτως ώστε οι νέοι να διδαχθούν το επιχειρηματικό πνεύμα. Να μην μαθαίνουν δηλαδή απλώς πώς να συμπληρώνουν αιτήσει για να προσληφθούν, αλλά να μαθαίνουν πώς πρέπει κανείς ε, να στήσει μια επιχείρηση και να την διοικήσει. Κύριε Μέντες Βάλτες, εσείς ε, έχετε μελέτες για να ε, εξακριβώσετε τις ανάγκες των επιχειρηματιών. Τι όργανα χρειάζονται για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Γιατί μαθαίνουμε ότι οι μικρομεσαίες ε, δημιουργούν όλο και λιγότερες θέσει εργασία. Άρα κάτι χρειάζεται να κάνουμε, χρειάζονται νέα μέσα. Μήπω πρέπει να τα ψάξουμε για να βρούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος. Μιχαέλα Ζιόντροβα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας για τις παρουσιάσεις τους και για το έργο που επιτελούν ε, οι φορείς τους. Έχω ασχοληθεί πολύ με εκθέσεις του ΣΕΝΤΕΦΟΠ και νομίζω ότι οι μελέτες αυτές είναι πολύ χρήσιμες για τις αποφάσεις που παίρνουμε στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και της αγοράς εργασίας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Εξέτασα το πρόγραμμα εργασιών σας για το 2016. Προτείνετε ορισμένες εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις, αλλά κάτι δεν το βλέπω εσείς που έχετε 40χρονη πείρα λειτουργίας υπέθετα ότι έχετε κάποιες ε, μακροπρόθεσμες ε, μελέτες συνολικής επισκόπησης. Οπότε κύριε Διευθυντά του ΣΕΝΤΕΦΟΠ, ποιες από τις μελέτες σας ε, έχουν ευρύτερο πρίσμα ή πρόκειται να εκπονήσετε τις μελέτες στο μέλλον. Για την κυρία Έρμπαν, Πέρυσι συζητούσαμε τη δυνατότητα ε, να έρθουμε σε επαφή με την Ουκρανία. Είχατε ορισμένα προγράμματα υποεκπώνηση για θέσεις μαθητείας στην Ουκρανία. Νομίζω ότι το αναφέρατε και την προηγούμενη φορά. Καταφέρατε να τα εφαρμόσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Χάβι Λόπεθ. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς και εγώ να ευχαριστήσω τους φορείς για την εργασία. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο για όλους τους θεσμούς και ειδικά για το Κοινοβούλιο. Αλλά να αναφερθώ σε κάτι που δεν αναφέρθηκε μέχρι τώρα γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την αγορά εργασίας. Αλλά το συζητάμε όλο και περισσότερο. Είναι κατανομή εισοδημάτων. Ξέρουμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες ανισότητες την κατανομή εισοδημάτων. Και έχει να κάνει πολύ βέβαια και με το γεγονό ότι η αμοιβή της εργασίας έχει μειωθεί και έχει αυξηθεί κατά πολύ η απόδοση του κεφαλαίου. Έχει αυξηθεί λοιπόν η ανισότητα στην κατανομή εισοδημάτων και κατά την κρίση διαπιστώσαμε ότι οι ανισότητες αυτές διαπιστώσαμε κατά την κρίση πέρα από την ηθική τους διάσταση ε, στρεβλώνουν και την ζήτηση και σε τελευταία ανάλυση θίγουν τους θεσμούς ε, και τη δημοκρατία. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ λέει Edith Bauer. Κύριε Χέντελ, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι πολύ που έχω τη δυνατότητα να ε, συμμετέχω σε αυτήν την οικία συζήτηση για τους οργανισμούς. Ακούγοντάς σας ε, θυμήθηκα τα συναισθήματα που είχα όταν ασχολούμασταν με τους οργανισμούς και μας ε, ε, είχαν πει ότι είμαστε πολύ τυχεροί ως επιτροπή που έχουμε να κάνουμε με αυτούς τους οργανισμούς σε σύγκριση με τους οργανισμούς με τους οποίους ασχολούνται άλλες επιτροπές πάντα. έχω μια συνολική θα έλεγα η εικόνα για τρεις τουλάχιστον από αυτούς τους οργανισμούς και το έργο τους. Και τώρα ως ε, αναπληρωματικό μέλος του Κοινοβουλίου στο ETF θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για όλους αυτούς τους οργανισμούς και ιδίως για το ETF. Το ETF διαφέρει σε έναν βαθμό από τους άλλους οργανισμούς και γιατί η σύνδεση του έργου του με την Επιτροπή μας δεν είναι τόσο στενή ή τόσο πρόβλη όσο στην ε, περίπτωση για παράδειγμα του οργανισμού του Δουβλίνου ή του Σεντεφόπ. Θα ήθελα λοιπόν να υπήρχαν πιο συνεκτικές και συντονισμένες πολιτικές. Γιατί, όπως μπορείτε να δείτε, το ETF θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό εργαλείο της, ε, πολιτικής, της αναπτυξιακής πολιτικής. Και ενδεχομένως ως Επιτροπή Απασχόλησης δεν ε, ε, ε, αξιοποιούμε πάντοτε επαρκώς αυτήν την ε, διάσταση. Και όπως είπε και η συνάδελφος, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας, ιδίως στις, σε νέες χώρες, θεωρώ ότι και μέσω του έργου του ETF θα μπορούσε να κατευθύνεται καλύτερα ε, προς και με αποδέκτη την εκπαίδευση και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ό,τι ε, συμβαίνει σήμερα. Αυτό δηλαδή που θα ήλπιζα να υπάρχει ε, θα ήταν ένας καλύτερος συντονισμός με την αναπτυξιακή πολιτική γιατί όπως είπα θα μπορούσε κάτι τέτοιο να αποτελέσει πολύ ισχυρό εργαλείο στον τομέα της μετανάστασης, στον τομέα της αναπτυξιακής πολιτικής και νομίζω ότι δεν κατευθύνουμε σε επαρκή βαθμό τις εμπειρίες που έχουμε συλλέξει ε, μέσα από τις πολιτικές μας προς τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Εγώ τέλος. Κάποια ερωτήματα θα θέσω, πολύ σύντομα. Συνδέονται όμως με αυτά που είπε και η Edith Bauer για, άλλους, ε, για άλλες επιτροπές. Ε, όταν ακούμε ότι οι οργανισμοί πρέπει να μειώσουν τον προπολογισμό τους, ε, τίθεται το ερώτημα, είναι καλό αυτό. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι κάτι καλό αυτό, ωστόσο είναι ένας στόχος. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαν τα αρνητικά αποτελέσματα αυτής της μείωσης να ε, αντισταθμιστούν μέσω μιας καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών ε, αυτών. Μεγάλη πρόκληση της για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η ε, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η ψηφιοποίηση όπως την ε, αποκαλούν άλλοι. Και πρόσφατα ρώτησα επίτροπο επί του θέματος και ε, η απάντηση ήταν ότι η τεχνολογική εξέλιξη πάντοτε φέρνει περισσότερη εργασία. Ήταν εθαρρυντική βεβαίως αυτή η απάντηση. Υπάρχουν μελέτες που ε, ε, σκεγραφούν πολύ θετικές προοπτικές ε, λόγω της ψηφιοποίησης, άλλες που καταλήγουν στα αντίθετα συμπεράσματα. Το ερώτημα μου είναι λοιπόν τι μπορεί να κάνει η Eurofound στο θέμα αυτό για να μας διαφωτίσει. Επίσης, όσον αφορά την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ένα, ένα ζήτημα που συζητείται διαρκώς είναι η κατάργηση ε, των ωραρίων εργασίας, το γεγονός ότι οι άνθρωποι ε, θα εργάζονται όλη τη μέρα, μέσα στη νύχτα. Ερώτημα για, προς τον James Καλέχα και ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα μαζί και είδαμε αυτό το, την έναρξη του προγράμματος μεταξύ Ελλάδας και Θουριγκίας... και ε, είδαμε ότι υπάρχει ε, εμπειρία και έχει διαπιστωθεί ότι οι δεξιότητες απέχουν πάρα πολύ από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τι μπορεί να κάνει το Σεντεφόπ για την αντιμετώπιση ε, αυτών των προβλημάτων. Και ένα τελευταίο ερώτημα για τη Ματλέν Σέρμπαν. Θεωρώ πολύ σημαντικά τα έργα που γίνονται σε άλλες χώρες. Όμως το ερώτημά μου είναι πώς σε αυτά τα έργα θα μπορούν να συμμετέχουν και η κοινωνική εταίροι. Τώρα, αν οι διερμηνείς μου δώσουν άλλα πέντε λεπτά, θα έχετε κι εσείς ε, λίγο περισσότερο χρόνο για να απαντήσετε. Δίνω το λόγο στην ε, κυρία Κρίστα Σέντλατσεκ. Ξεκινώ με το πρώτο ερώτημα. Της κυρίας Στάινρουκ, γι' αυτό και θα απαντήσω στα γερμανικά. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και τι συμβαίνει ε, με την υποστήριξη αυτών των επιχειρήσεων και τι μπορεί να κάνει ο οργανισμός μας. Εμείς έχουμε δύο βασικές δραστηριότητες. Τη μία την ανέφερε που είναι αυτό το ΟΙΡΑ, το εργαλείο αξιολόγησης κινδύνου που βοηθά ε, την ε, αξιολόγηση του κινδύνου από τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Βλέπουμε και το απέδειξε και η μελέτη ότι τα τελευταία χρόνια το εργαλείο αυτό χρησιμοποιήθηκε από πολλές μικρές επιχειρήσεις σε πολλούς κλάδους ότι η κοινότητα των χρηστών διευρύνεται διαρκώς και είναι ένα παράδειγμα για το πώς εμείς οι οργανισμοί μπορούμε τελικά να επηρεάσουμε θετικά το έργο των επιχειρήσεων και όσον αφορά την ε, στρατηγική ε, για την προστασία στην εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρώ ότι κινούμαστε στην σωστή ε, κατεύθυνση περισσότερες πληροφορίες για το τι χρειάζονται αυτές οι επιχειρήσεις θα μας προσφέρει και η νέα έρευνα για το τι γίνεται για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και μετά το επόμενο ερώτημα για το στρες στον χώρο εργασίας. και τη διάσταση του στρες από τον εξωτερικό κόσμο, που προέρχεται από τον εξωτερικό κόσμο. Ναι, βλέπουμε ότι στην εκστρατεία μας, σε όλα τα κράτη-μέλη και σε επίπεδο εταιρεία βλέπει κανείς ότι υπάρχει πάντοτε ένα μείγμα ε, ψυχοκοινωνικών κινδύνων σε επίπεδο εταιρεία, αλλά υπάρχουν και πηγές στρες από τον εξωτερικό κόσμο. Εμείς επικεντρωνόμαστε στην ευθύνη των εργοδοτών και των εταιριών να βοηθούν τους εργαζόμενούς τους να αντιμετωπίζουν το στρες και να λαμβάνουν μέτρα για να βοηθούνται οι εργαζόμενοι. Διαχείριση ε, στρες βεβαίως σημαίνει να μειωθεί το στρες και στο χώρο εργασίας αλλά και ε, η χρήση εργαλείων όπως η ε, πρόληψη. Χρειάζεται δηλαδή ορισμένες φορές και κάποια εξωτερική βοήθεια από ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ιδιωτική τους ζωή. Άρα φυσικά ε, επικεντρωνόμαστε περισσότερο στο επίπεδο της εταιρείας, των εταιριών και βλέπουμε ότι το ε, στρες αυξάνεται εκεί Παρ' όλα αυτά, οι εργοδότες έχουν στα χέρια τους μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να μειωθεί το στρες, μεταξύ άλλων και μέσω της καλύτερης οργάνωσης των δραστηριοτήτων. Τέλος, αναφέρθηκε ότι Έχουμε δραστηριότητες που αντιμετωπίζουν ή απαντούν λίγο ή πολύ στο, στα ίδια ζητήματα. Την αγορά εργασίας. Εμείς στον όσα συνεργαζόμαστε στενά με τη Eurofound και τώρα και με το Σεντεφόπ για παράδειγμα στη νέα εκστρατεία για τον γυράσκοντα ε, εργαζόμενο πληθυσμό Θέλω να πω όμως ότι εμείς έχουμε συμπληρωματικό ρόλο ως προς το έργο μας, δηλαδή αξιοποιούμε το έργο και της Eurofound και της Sendefop ε, και βεβαίως λαμβάνουμε υπόψη τα απορίσματα στα οποία έχουν καταλήξει όλοι οι οργανισμοί που ε, ασχολούνται με την αγορά εργασίας. Η υγεία Είναι πράγματι σημαντικό θέμα. Δεν το αναγνώρισαν κάποιες χώρες έγκαιρα. Αν θέλουμε όμως οι άνθρωποι να παραμένουν υγιείς έως τη συνταξιοδότηση τους θα πρέπει να καταβληθούν πολύ περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Όπως ανέφερα, το διετές πρόγραμμα για τους ηλικιωμένους εργαζόμενούς μας κατέδειξε σαφώς ότι υπάρχει ανάγκη να ε, υπάρξουν βελτιώσεις και να ληφθούν μέτρα σε πολλά επίπεδα. Υπάρχει το επίπεδο της πολιτικής όπου θα πρέπει να εκπονηθούν, να συνταχθούν στρατηγικές για τη βελτίωση της κατάστασης και να αναπτυχθούν στρατηγικές ή ε, συστήματα παροχής βοήθειας προς τις εταιρείε, αλλά υπάρχει και το επίπεδο των εταιριών οι οποίες από την πλευρά τους θα πρέπει να λάβουν μέτρα και να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Και θα παρουσιάσουμε τα προορίσματά μας αυτά πολύ σύντομα γιατί ε, εμείς ε, αναλύσαμε τέσσερις ομάδες χωρών στην Ευρώπη και η κάθε από αυτές τις ομάδες ε, αντιμετωπίζει τα προβλήματα στον χώρο εργασίας με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν κάποιες χώρες, μια ομάδα χωρών η οποία είναι και η καλύτερη να το πω έτσι, που άρχισε να ε, αντιμετωπίζει πιο έγκαιρα, έγκαιρα από τις άλλες τα προβλήματα αυτά. Δυστυχώς πρέπει να σταματήσω. Ξαφνικά έκλεισε η φωνή μου. Με συγχωρείτε. Κύριε Καλέχα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Με ενθαρρύνει πολύ το ότι εσείς που βρίσκεστε ε, στο μέτωπο λέτε σε εμά που βρισκόμαστε από πίσω τι πραγματικά συμβαίνει στην κοινωνία. Οι ερωτήσει λοιπόν που κάνετε είναι πολύ σημαντικέ για εμά ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα του 16, του 17, του 20 θα κινηθούν προ την κατεύθυνση στο σχολείο του Προέδρου ε, για το ζήτημα των περικοπών. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι όλοι οι οργανισμοί μαζί και ε, διορθώστε με αν κάνω λάθος χρησιμοποιούν το 2% και λιγότερο του συνολικού προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λοιπόν φωνάζουμε για περισσότερα είναι αυτό απόλυτα αιτιολογημένο αν δει κανείς ε, πόσο πολυάριθμα είναι τα ζητήματα που θίξατε. Χρειαζόμαστε νέα κονδύλια και περισσότερους πόρους. Τώρα όσον αφορά τα προγράμματα μαθητία. Εμεί ξεκινήσαμε τι αναθεωρήσει, είναι πολύ επιτυχη. Πολύ ενθαρρυντικά τα στοιχεία όταν συζητούν μεταξύ του οι κοινωνικοί εταίροι για τόσο βασικά ζητήματα όπου πρέπει να συναντώνται η εκπαίδευση και η απασχόληση. Έχουμε την εμπειρία στη Λιθουανία, στην Μάλτα, στην Ιταλία και στη Σλοβενία και στην Ελλάδα ειδικότερα. Όπου, όπω είπε ο πρόεδρο, όταν μιλάμε για επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, η απόσταση μεταξύ αυτή τη κατάρτιση και τη αγορά εργασία είναι ε, τεράστια. Εκεί πρέπει να χτίσουμε γέφυρες. Ε, όσον αφορά του πρόσφυγες και τι σχετικέ μελέτε, πέρυσι ε, δημιουργήσαμε μια ομάδα εργασία τη ΕΔΕΦΟΠ για να χαράξουμε την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η ΣΕΔΕΦΟΠ τουλάχιστον το 2017 με ένα σχέδιο δράση ώστε να βρει έναν τρόπο να βοηθήσει τα κράτη-μέλη για το ζήτημα των προσφύγων. Σκοπημένο είναι να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι το Δεκέμβριο η Κομισιόν και εμείς δημοσιεύσαμε τις ευρωπαϊκές καθημερινές γραμμές για την επικύρωση της άτυπης και μη τυπικής ε, μάθησης. Η δημιουργία προφίλ για τους πρόσφυγες ε, πρέπει να έχει προτεραιότητα. Ποιοι είναι αυτοί οι πρόσφυγες, τι ικανότητες και δεξιότητες έχουν, πώς μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, τι άλλες δεξιότητες χρειάζονται. Και φυσικά η πρώτη δεξιότητα θα είναι οι γλώσσες, οι ικανότητες, η συμπεριφορά, ε, δεξιότητες που σχετίζονται με την πληροφορική. Υπάρχει ποικιλία ζητημάτων που εξακολουθούν να μας είναι ασαφή όσον αφορά το τι θα χρειαστούν οι πρόσφυγες για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητά μας όπως ξέρετε υπάρχουν εργαλεία δημιουργίας προφίλ ε, στην ε, Σουηδία και στη Γερμανία και εμείς σκοπεύουμε να κάνουμε μια συνάντηση με αυτές τις δύο χώρες για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εφόσον υπάρχουν ήδη εργαλεία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το Europass, όπως το Ευρωπαϊκό Πανόραμα Δεξιοτήτων που ξεκινήσαμε πέρυσι και κατευθείας γραμμές για την επικύρωση, όλα αυτά τα εργαλεία δεν μπορούμε να τα αφήσουμε σε μια βιβλιοθήκη ούτε πάνω σε ένα τραπάζι. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε στην πρακτική. Όταν υπάρχει συνέργεια μεταξύ των οργανισμών μας, ενημερωτικά, ε, μοιραζόμαστε γνώση μεταξύ μας μέσω σεμινωρίων και κάποιος αναφέρθηκε στην έρευνα εταιριών, η Κρίστα αναφέρθηκε σε μια άλλη δραστηριότητα που οργανώνουμε μαζί. Ε, τέτοιε δραστηριότητες κάνουμε δύο φορές το χρόνο και κοινοποιούμε ένα στον άλλο τα προγράμματα εργασιών μας ακόμα και για τα 17-20 ώστε να υπάρξει συνέργεια μεταξύ μας για τις διάφορες δραστηριότητε. Τώρα το ζήτημα των ατόμων εκτός εκπαίδευση απασχόλησης ή κατάρτισης τον ενητη 12% για τις ηλικίες 15 και 24 και 16% για τις ηλικίες 18 έως 24. Η αντίστοιχη της εκπαίδευσης με την απασχόληση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις ΕΝΤΕΦΟΠ. Το να φέρουμε αυτά τα δύο πράγματα πιο κοντά. Το να μάθουμε από τις εκμάθησεις μέσω των εταιριών είναι κάτι που ξεκινήσαμε πέρυσι. Ονομάζεται Learning Cultures and Organizations. Ε, κοιτάμε τι συμβαίνει στις ε, επιχειρήσεις για να το αντιγράψουμε στις, ε, ε, στην παιδεία και να δούμε πώς μπορεί αυτό να μεταφερθεί και σε άλλες επιχειρήσεις για τις μαθητείες. Θα ξεκινήσουμε το πίνακα βαθμολογίας για την κινητικότητα, όχι για να βαθμολογήσουμε χώρες και να τις ταξινομήσουμε ή να τι κάνουμε να φάνουν ανταγωνιστικές. Απλά βοηθάμε τα κράτη-μέλη να προσφέρουν υψηλότερη ποιότητα κατάρτιση και εκπαίδευση, ώστε και μαθητευόμενοι και εκπαιδευτέ να μπορούν να κινηθούν ελεύθερα εντό και εκτό των χωρών του. Φυσικέ συμβουλέ που δίνουμε στου νέου όσον αφορά τι δεξιότητε, ε, κάτι που ρωτήθηκε επίση. Εμεί ε, υπογραμμίζουμε το ζήτημα των γλωσσών, των μαθηματικών, των τεχνολογιών, τη πληροφορική, τη επιχειρηματικότητα και κυρίω κατά πόσο η εκάστοτε δεξιότητα μπορεί να, ε, και η, οποία μπορεί να, ε, δεξιότητα τη ε, συμπεριφορά, τη καλής συμπεριφοράς που μπορεί να μεταφερθεί στην αγορά εργασία. Όλο, ξέρετε, και περισσότεροι επιχειρηματίε έρχονται στη ΣΕΔΕΦΟ από ό,τι παλιότερα. Έχουμε ανοιχτεί προ τον ιδιωτικό τομέα, από τον οποίο θέλουμε να μάθουμε πράγματα, γιατί ξέρουμε ότι ο ιδιωτικό τομέα δημιουργεί θέσει εργασία. Και πρέπει λοιπόν να συμμετέχει απόλυτα στις δικέ μα πολιτικέ δημιουργίε θέσεων εργασία επισκόψη των μελετών που κάνουμε εδώ και χρόνια στη ΣΕΝΤΕΦΟΠ έχουμε διαδικασία της Κοπενχάγης πρώτον που ξεκίνησε το 2002 και συνεχίζει να είναι ένα συνεχόμενο έργο μας έχει μεταφερθεί στα παρατέρα της Μπρούς και μετά της Ρήγας όλο ένα αυξάνεται δηλαδή και μετά έχουμε και τα ευρωπαϊκά εργαλεία που αποτελούν βασική πτυχή της εργασίας μας Αυτά θα καθορίσουν το μέλλον της κινητικότητας μεταξύ των κρατών μελών, αν θα συνεχίσει να υπάρχει όχι. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες σας ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, James Καγιάχα. Παρακαλώ δώστε μας ε, μερικά λεπτά ακόμη από τη ε, να απαντήσει η κυρία Σαρβάν και μετά τελειώνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις που μας βοηθάνε και στο έργο μας. Θα ξεκινήσω με τον εκδημοκρατισμό. Σας ευχαριστώ πολύ και για τις ευχαριστίες που αποστήλατε στο προσωπικό μας. Και είμαι εδώ και με εκπρόσωπο του προσωπικού του οργανισμού μας ETF. Και νομίζω ότι είναι σωστό που έχουμε αυτή τη συνεργασία τη δημοκρατία, τη δημοκρατία τη θεωρούμε κάτι το αυτονόητο στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι αυτονόητη στις γειτονικέ μας χώρες. Εάν δεν υπάρχει η σωστή κατάρτιση για τη σωστή διακυβέρνηση, αν δεν προωθήσουμε μία ε, προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς με τη συμμετοχή των ε, τοπικών αρχών, του ιδιωτικού τομέα, εάν όλοι αυτοί ε, συναντιόνται και μάλιστα όχι τυπικά αλλά ουσιαστικά, τότε μόνο θα επιτύχουμε. Η εργασία μας λοιπόν είναι να τους βοηθήσει να προσεγγίσουν ο ένας τον άλλον και να γίνουν αξιόπιστοι εταίροι. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις. Υπάρχει κάποιος εκδημοκρατισμός από πλευρά των εργοδοτών, αλλά χρειαζόμαστε πολύ στήριξη από τα κράτη-μέλη όταν εργαζόμεθα με τα συνδικάτα σε σχέση με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Αυτό δεν είναι τόσο ανεπτυγμένο στι χώρε με τι οποίε συνεργαζόμεθα, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων χωρών. Τώρα, για την εκπαίδευση ε, στην επιχειρηματικότητα. Βεβαίω, είναι βασικό στοιχείο, είναι τμήμα ε, των προσπαθειών που κάνουμε παντού για να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών. Σε όλες τις χώρες, στην Νότια Μεσόγειο για παράδειγμα, στο Λίβανο για παράδειγμα ε, είναι περισσότερο πρόθυμοι γιατί είναι στο γονιδίωμά τους και το κάνουμε και στην Ιορδανία, στην Τινησία, το Μαρόκο αλλά δεν θέλουμε απλώς να μπει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να εκπαιδεύσεις και τους ε, καθηγητές Πρέπει να είναι σωστά εκπαιδευμένοι οι καθηγητές, να έχουν τη σωστή στάση, να είναι διατεθειμένοι να λαμβάνουν κινδύνους, να ψάχνουν για λύσεις. Και απευθυνόμεθα και προς τους νέου επιχειρηματίε και τις γυναίκες επιχειρηματίε. Στην Ευρώπη θεωρούμε ότι η συμμετοχή των γυναικών είναι επίση αυτονόητη. Αλλά πριν από 50 χρόνια, για παράδειγμα, ιδιαίτερα στι χώρε μα η συμμετοχή των γυναικών στην εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα ήταν πολύ χαμηλή και σε ορισμένε ακόμη πρέπει να γίνουν πολλά και πρέπει να εστιάσουμε και σε αυτό στο εγγύ μέλλον. Τώρα για τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε είναι σε κατάρτιση. Του λεγόμενου needs. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση γι' αυτό. Βεβαίω είναι πολύ σημαντικό θέμα. Από τα πιο σημαντικά. Γιατί έχουμε 2,8 εκατομμύρια νέου. Στη Συρία για παράδειγμα. Που είναι ακριβώ σε αυτή την κατάσταση και έχουν περιορισμένες δυνατότητες ε, να επιτύχουν κάτι. Και η Συρία είναι μία από τις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμεθα. Και αν δούμε είναι μία από τις πρώτες περιόδους που εργαζόμεθα εκτός Ευρώπης. Και προσπαθείς να καταλάβεις πώς σχετίζεται με τη ριζοσπαστικοποίηση και τρομοκρατία. Είναι προφανές ότι σχετίζεται και υπάρχει κίνδυνος ε, Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε πολύ περισσότερο για να τους δώσουμε κάποια προοπτική. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σε ορισμένε από αυτέ τι χώρε μαζί με τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, και δεν θα συζητήσω τώρα γι' αυτό, με βάση τις θετικέ ε, εμπειρίε που έχουμε από την εργασία με τους Παλαιστίνου πρόσφυγες έχουμε λοιπόν πολλά να κάνουμε. Επίσης υπάρχουν πρόσφυγες και στις χώρες εταίρους μας ε, Τουρκία, Λίβανος, Ιορδανία, πρέπει να κάνουμε πολλά και σε αυτές τις χώρες. Και σας ευχαριστώ και για την ερώτηση για την Ουκρανία. Α, και με εντυπωσιάζει το ότι θυμάστε αυτά που είπαμε πέρσι. Ναι, κάναμε την εξάντε μελέτη αντικτύπου για τη βελτίωση της παρέμβασής μας στα σχολεία και ε, μας έχει εντυπωσιάσει ότι όλες οι περιφέρειες, υπογραμμίζω όλες οι περιφέρειες της Ουκρανίας εργάζονται για να διασφαλίσουν αυτήν την αντιστοίχηση δεξιοτήτων και αναγκών στην αγορά εργασίας. Δεν θα μιλήσω τώρα για τις περικοπές. Ε, ελπίζω ότι θα μας βοηθήσετε, θα μας δώσετε περισσότερες πιστώσεις και ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο Χάν Μενέντες Βάλτες. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω από την ε, ψηφιακή μετάβαση και την τέταρτη επανάσταση που αναφέρατε στην τελευταία σας παρατήρηση. Που φτάνουμε σε κάτι που είχε προβλεφθεί πολλάκις και πάντα ήταν λάθος η πρόβλεψη αλλά τα πράγματα τώρα έχουν αλλάξει. Παρακολουθούμε τις διαφορετικές αλλαγές και η δημιουργία αυτού του χάσματος μεταξύ εργασιών και εκπαίδευσης ε, ανάμεσα σε δύο άκρα σχετίζεται με τη δυνατότητα αντικατάστασης ορισμένων κλασικών δραστηριοτήτων. Αυτό είναι μέρος της εξήγηση. όχι μόνο τώρα με τις νέες τεχνολογίες. Ε, όμως δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε μόνο καθημερινές εργασίες, αλλά και οτιδήποτε είναι προβλέψιμο, ότι λειτουργεί βάση μοτίβου, οπότε υπάρχει η δυνατότητα. Τώρα η έκταση δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι όχι μόνο θα αλλάξουν οι διαθέσιμες εργασίες, αλλά και η μορφή του κόσμου όπως το ξέρουμε. Η τόποι εργασία μας, οι ώρες εργασίας μας, η σχέση μας με τους εργοδότες, ε, το κατά πόσο θα κάνουμε μια ολοκληρωμένη εργασία ή ένα μέρος της μόνο κτλ. κτλ. Οπότε τέτοια ερώτηση τι χρειάζεται, τι μπορούμε να προβλέψουμε για το μέλλον. Πραγματικά δεν ξέρουμε. Σε τελική αναλύση είναι η δυνατότητα διαρκούς προσαρμογής και οι εφαρμόσιμες ε, δεξιότητες είναι ένας σημαντικός παράγοντας ε, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων που δεν σχετίζεται με κάποια τεχνική απέτηση ε, κάποιου συγκεκριμένο τομέα. Τώρα η κυρία Στάινμπροκ ρώτησε για την ποιότητα των θέσεων εργασία. Ναι, εμεί παρακολουθούμε την εξέλιξη της ποιότητας εργασίας εδώ και 25 χρόνια. Αλλά μπορεί οι αλλαγές να φέρουν μια άλλη εικόνα, διότι τα συμπεράσματά μας είναι ότι τα τελευταία χρόνια τα πράγματα είναι σχετικά σταθερά. Κάποια πράγματα βελτιώνται, αλλά όχι ή επιδηλώνονται λίγο και μας ανησυχούν. Αυτό οφείλεται εν μέρη στον αριθμό των θέσεων εργασίας που είναι διαθέσιμες, αλλά η εικόνα που έχουμε διαμορφώσει εμείς είναι ότι στην Ευρώπη έχουμε εργαζομένους ε, αφενός ε, που ενθαρρύνονται από τον οργανισμό από τους συναδέρφους τους που είναι ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους όπου υπάρχουν περισσότερες γυναίκες ε, προϊστάμενοι κτλ. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν και κάποια αρνητικές επιπτώσεις, πίεση που επηρεάζει την κοινωνική συμπεριφορά που μπορεί να επηρεάσει ε, ουσιαστικά όλο και μεγαλύτερη ένταση στο χώρο εργασία που δεν συνοδεύεται από αυξημένη αυτονομία. Ο διαρκής διαχωρισμός των φύλων στην αγορά εργασίας, ο αριθμός των ωρών εργασία που είναι υψηλότερος για τις γυναίκες εάν υπολογιστεί όχι μόνο ο αμοιβόμενος χρόνος εργασίας, αλλά και ο μη αμοιβόμενο. Θα δείτε κάποιες πληροφορίε στα πρώτα ευρήματα που έχουμε δημοσιεύσει. Τώρα όσον αφορά την κατάσταση που ανέφερε η Τζούδιθ και οι άλλοι συναδέλφοι. Συνεχίζουμε το έργο μας ε, για τους ε, ανθρώπους εκτός απασχόλησης, και εκπαίδευσης. Το θέμα εκεί είναι να ξεμπλέξουμε τις διάφορες ομάδες, να ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι ποιες. Κάποιες ε, δημιουργούν περισσότερες ανησυχίες από άλλες. Φέτος, ας πούμε, θέλουμε να εστιαστούμε στους πολύ μακροχρόνια νέους ανέργους αλλά επίση είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη και η κατηγορία των ανθρώπων που έχουν αποθαρρυνθεί και έχουν μείνει αδρανεί. Είναι η πιο δύσκολη κατηγορία και διάφορε αξιολογήσει λένε ότι οι διάφορε πολιτικέ δεν φέρνουν πάντα αποτέλεσμα. Έχουμε συμβάλει σε κάποιε αξιολογήσει ε, και έχουμε υποστηρίξει και το ελεγκτικό συνέδριο σε κάποιου ελέγχου επιδόσεων σε επίπεδο κρατών μελών για την υλοποίηση τη εγγύηση για του νέου βάσει των ευρημάτων αυτών. Λοιπόν, ε, και τώρα αναφερόμενο στο δικό μας προσωπικό, ξέρετε, να τονίσω είναι πολύ σημαντική η έμπρες του προσωπικού μας. Τώρα η αντιστοιχεία των δεξιοτήτων και η κινητικότητα, το 40% των εργοδοτών λένε ότι δεν βρίσκουν ανθρώπους σωστά καταρτισμένους ακόμα και σε χώρες με υψηλή κατάρτιση, με υψηλή ε, απασχόληση. Θέλουμε λοιπόν πραγματικά να προωθήσουμε την κινητικότητα ή θέλουμε να την ε, σταματήσουμε. Αυτό συζητείται αυτή τη στιγμή. Δεν έχει και μεγάλη υποστήριξη κινητικότητα ακόμα και εντός κρατών μελών. Παρότι θεωρητικά θεωρούμε ότι περισσότερα έχει να κερδίσει κανείς παρά να χάσει. Τώρα για τους εργοδότες, και εδώ θα κλείσω, κάναμε μια έρευνα σε εταιρείε όπου λέγεται η ότι είναι σημαντικό να παρέχουμε και κάποιες προφορίες για τις επιχειρήσεις, για το management τους, ε, ε, τις επιχειρήσεις που κάνουν καλύτερη δουλειά στη δημιουργία θέσεων εργασία. Να ε, τελειώσω με την κατανομή εισοδήματος στον κύριο Λόπες και θα απαντήσω στα ισπανικά. Σίγουρα η κατανομή εισοδημάτων και αποδοχών είναι κάτι που το μελετήσαμε και φέτος τώρα ολοκληρώνουμε μία μελέτη γενικότερα για την κατανομή εισοδημάτων υπάρχουν ανισότητες. Ε, Βέβαια δεν είναι μεγαλύτερες από τις ανισορροπίες που διαπιστώνουμε, τις ανισότητες που διαπιστώνουμε στις Πολιτείες. Αλλά έχει υπάρξει ε, αύξηση αυτών των ανισοτήτων σε σχέση με την προκρισιακή περιοχή, ε, περίοδο. Δεν έχω χρόνο, θα μπορούσα ώρες να τα λέω, αλλά... Και εμείς θα μπορούσαμε να καθίσουμε ώρες να σας ακούμε. Αλλά θα πω μόνο ότι το έργο σας είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τη δική μας επιτροπή, για να αναφερθώ και στην παρέμβαση της Edith Bauer. Δεν χρειάζεται όμως να το πω αυτό. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Θα ήθελα επίσης να μεταφέρετε τους χαιρετισμού μας μέρους της Επιτροπής στους εργαζόμενους των οργανισμών σας για το έργο τους. Και φυσικά οι προκλήσεις θα μεγαλώνουν όσον αφορά και τις ε, μελλοντικέ εξελίξεις πολιτικά και οικονομικά. Κάτι που θα ε, διαπιστώσουμε και στην ε, διαδικασία της ψηφιοποίησης οικονομίας και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να βασιζόμαστε στο έργο σας γιατί οι οργανισμοί μας είναι και όταν λέω μας, εννοώ δεν θέλω να, ε, ε, το λέω γιατί δεν θέλω να ιδιωτικοποιηθούν. Γιατί μπορούμε εμείς να συμμετέχουμε στο έργο το δικό σας, να το συνδράμουμε, αν το χρειάζεστε, αν θέλετε εσείς μια τέτοια στήριξη, εμείς είμαστε στη διάθεσή σας και με τη γραμματεία μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας εδώ. Θεωρώ ότι θα τα πούμε πολύ σύνταμα και πάλι. Να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς και για το λίγο χρόνο παραπάνω που μας διέθεσαν και θα τα ξαναπούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής μας στις 16 και 17 Μαρτίου. Καλή σας μέρα.